Καλημέρα σα. Καλώ ορίσατε. Θερμά. Συνεχίζεται η συνεδρίασή μα, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχά, αποφάσει των συντονιστών των δύο τελευταίων συνεδριάσεων τη 7 η Απριλίου και χτεσινή ε, σα διανέμονται τα αντίγραφα, δεν έχετε αντιρρήσει μέχρι το 12.30 σήμερα το μεσημέρι θα θεωρηθούν εγκεκριμένε οι αποφάσεις. Πάμε στη ψηφοφορία για τη συμφωνία ε, με τα Ηνωμένα Έθνη για τα άτομα με αναπηρία. Ο κύριο Κέλετς είναι ο νομοδότηση. νομοδότησης. Εμείς νομοδοτούμε στην Επιτροπή ΕΜΠΛ ε, απασχόλησης. Άρχεται η ψηφοφορία, είναι δοκιμαστική αυτή για να δούμε τα μηχανήματα παρακαλώ. πέρας, όχι και πέρας, είπα και εγώ όπως είσαστε ε, ακριβώς. <laughs> εντάξει, εντάξει, τώρα είναι όλα καλά. Ψηφίζουμε. Τροπολογία παριθμών 12. Ψηφί πέρα, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 13 πέρα κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 19. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Υπέρ. Υπέρ. Καταπίπτει λέει ο κύριος Βαντεκάμπ. Α, εγκρίθηκε η 17 μάλιστα. Οπότε καταπίπτει. Μα, όχι, απερίφθη 17. Βιμ Βαντενκάμπ, εντάξει κατάλαβες. Λοιπόν, το τμήμα 1 της 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές, αυτό θέλει έλεγχο. Το δεύτερο τμήμα της 19 άρχεται ψηφοφορία τώρα. Πέρασε.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 κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οπότε πηγαίνουμε στην 35 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 49 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τσεκ φωνές. Την 49 την ελέγχουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Abstimmung ist geschlossen. 25 ε, υπέρ 16 κατά μία αποχή. Χρειάστηκε όλα έλεγχος, πραγματικά χρειαζόταν. Ε, πού είχαμε μείνει τώρα. Στην 51. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Την 61 παρακαλώ τσεκάρουμε αρχίζει τώρα ηλεκτρονική απολύθευση. πέρας 18 υπέρ 25 κατά χωρίς αποχές. Απορρίπτεται. 62 Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παρθών 1 υπέρ. Κατά.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 Αρχίζει. Και τελειώνει. Με μία ψήφο κατά, 41 υπέρ, μία αποχή. Συν μία υπέρ, χωρίς κάρτα, 42. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια ε, στον κύριο Σκρέλιτς.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 Ερχόμαστε τώρα στην παρουσίαση της έκθεσης με τις συστάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου ε, για τις εμπόλεμες περιοχές. Ξέρετε, αυτό έγινε μετά την τραγική κατάρριψη ε, του αεροσκάφους Boeing 777 των Μαλισιανών αερογραμμών τον Ιούλιο του 2014. Μετά από εγκληματική εκτόξευση ρουκέτας έχασαν τη ζωή τους 298 άνθρωποι και πολλοί κατάγονται από τις κάτω χώρες. Το Νοέμβριο της ε, το 2015 μας παρουσίασε ο αντιπρόεδρος ε, της ε, Ολλανδικής Υποεπιτροπής για την Ασφάλεια τα αποτελέσματα και τα πορίσματα ε, της έκθεσης. Ο κύριος Κι ήταν παρόν και αναφέρθηκε τότε το θέμα των αδυναμιών και των προβλημάτων των εθνικών συστημάτων. Περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία να ακούσουμε τα απορίσματα και τα συμπεράσματα της δικής σας μελέτης. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι ευρωβουλευτέ, είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα αυτή τη σημαντική ειδική ομάδα. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε, όπως αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, ως αποτέλεσμα του τραγικού γεγονότος που ε, συνέβη στην Ουκρανία το 2015. και προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε τι χρειάζεται να γίνει από ευρωπαϊκής πλευράς για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που υπάρχει. Γνωρίζοντας ότι δυστυχώς ο κόσμος δεν είναι πιο ασφαλής ε, τώρα πια από ό,τι στο παρελθόν και ότι μπορεί να υπάρξουν ε, απειλές ανάλογες ε, με αυτό που συνέβη στην Ουκρανία. Η ειδική ομάδα εργάστηκε επί τρεις μήνες. Η τελική έκθεση δόθηκε στην Επίτροπο Μπούλ στον Μάρτιο και εστάλει και στην Ολλανδική Προεδρία για να ληφθεί υπόψη στις εργασίες του Συμβουλίου για την αναθεώρηση του βασικού κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Έχετε όμως και εσείς την ευκαιρία να εξετάσετε την έκθεση και τις συστάσεις ε, του Ολλανδικού Φορέα. Στην ειδική ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, της Γενικής Διεύθυνσης MOVE και HOME, από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ιδιαίτερα από το στρατιωτικό προσωπικό καθώς επίσης από το Κέντρο Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε εκπροσώπους ε, των κρατών μελών επίσης και πολύ ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τις ε, αρχές πολιτικής ε, αεροπορίας, αλλά είχαμε και εκπροσώπους του κλάδου. Επίσης είχαμε από την ΕΑΣΑ εκπρόσωπο και επίσης ε, είχαμε πρόεδρο ε, από την ΙΚΑΟ, η οποία έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Τι συζητήσαμε και τι διαπιστώσαμε. Καταρχάς, ε, διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση στα κράτη-μέλη διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και μάλιστα πολύ λίγα κράτη-μέλη έχουν πρόσβαση σε στρατιωτικές πληροφορίες όσον αφορά την απειλή. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ειδικέ ομάδε που συνεργάζονται στενά με τι ε, αρχέ πολιτική αεροπορία ε, αλλά και με τι ε, στρατιωτικέ υπηρεσίε πληροφοριών και γενικά με τι υπηρεσίες υπηρεσίε πληροφοριών. Αυτό όμω δεν συμβαίνει στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρώπης, όπου οι αρχές πολιτικής αεροπορίας δεν έχουν πρόσβαση σε στρατιωτικές πληροφορίες. Διαπιστώσαμε επίσης ότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη την δυνατότητα να εμποδίσουν τις δικές τους αεροπορικές γραμμές να ακολουθήσουν μια επικίνδυνη διαδρομή. Κάποια κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα αυτή, ιδιαίτερα αυτά που έχουν ομάδες αξιολόγησης κινδύνου και πρόσβαση στις στρατιωτικές πληροφορίες, αλλά τα περισσότερα άλλα κράτη-μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. και βασίζονται ε, σε, στο να τους πει κάποιος ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός ε, για να κινητοποιηθούν. Στην ομάδα μας είχαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με την έννοια των εθνικών αεροπορικών γραμμών και και ε, οι διάφορες αεροπορικές γραμμές αντιμετωπίζουν διαφορετικούς κινδύνους. Ε, στο παρελθόν είδαμε τρομοκρατικές ε, πράξεις που είχαν στόχο συγκεκριμένη εθνικότητα. Τώρα όμως που έχουμε ενιαία αγορά στην αεροπορία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πια αυτός ο όρος των εθνικών αερογραμμών και όπως αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, στην ε, πτήση των ε, αερογραμμών της Μαλαισίας οι περισσότεροι ε, επιβάτες ήταν Ολλανδοί. Διότι με τους κοινού κωδικούς πτήσεων μπορεί κανείς να αγοράσει ένα ειστήριο από Ολλανδική εταιρεία αλλά να βρεθεί σε αεροπλάνο των Μαλαισιανών αερογραμμών. Είναι λοιπόν κάπως ασαφής ο όρος αυτός των εθνικών αερογραμμών και Τούτου λεχθέντος θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, οι British Airways, η Air France και η Lufthansa αντιμετωπίζουν κάπως διαφορετικό κίνδυνο από αυτόν που αντιμετωπίζουν αεροπορικές εταιρείες από άλλες χώρες. Λόγω ε, της ε, συμμετοχής των χωρών αυτών σε διάφορες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Εάν όμως έχω πληροφορίες για κάποιον κίνδυνο, ο κίνδυνος αυτός αφορά μια χώρα, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά τους επιβάτες ε, και πώς ε, θα χειριστούμε τον κίνδυνο αυτόν. Και το συμπέρασμά μας ήταν να πούμε ότι αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες εταιρείες ε, που αντιμετωπίζουν ε, αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με άλλες. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο ε, κινδύνου το οποίο αφορά όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτόν τον κίνδυνο θα πρέπει να ασχοληθούμε και να αντιμετωπίσουμε. Επίσης διαπιστώσαμε ότι κάποιες φορές πρέπει να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. το τελευταίο δίμηνο. Είχαμε κάποια μηνύματα σχετικά με δοκιμές ε, πυράβλων στο Ιράν. Οι υπερπτήσεις του Ιράν γενικά δεν θεωρούνται επικίνδυνες, ωστόσο είχαμε δοκιμές βαλιστικών πυράβλων χωρίς προειδοποίηση στην διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα τις αρχές ε, ε, πολιτικής αεροπορίας. Τι θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε, να ε, έρθουμε σε επαφή με τις Ιρανικές αρχές και πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, μέρες, ώρες, νομίζω ώρες έως και λεπτά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα θέματα που συζητήσαμε λοιπόν ε, στην ειδική ομάδα ήταν μπορούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν ε, για να έχουμε ε, κοινή αξιολόγηση κινδύνου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως μέχρι τώρα, δηλαδή κάθε χώρα να εργάζεται ξεχωριστά. Η δεύτερη ερώτηση ήταν ποιος θα διαδίδει τις πληροφορίες για τον κίνδυνο που υπάρχει και πώς. Πολύ σημαντική ερώτηση. Ποιο ευθύνεται γιατί σε περίπτωση ατυχήματος ε, Κάποιο γνώριζε τον κίνδυνο, οι πληροφορίες αυτές είτε διαβιβάστηκαν είτε όχι, ποιο είναι υπεύθυνος για το τι έγινε με τις πληροφορίες αυτές. Και τέλος, μπορούμε να καθορίσουμε μια διαδικασία ε, για επίγουσες καταστάσεις. Είναι πολύπλοκη η εικόνα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Οι αρχές όμως ε, είναι πολύ απλές. Καταρχάς υπήρχε συμφωνία εντός της ειδική ομάδας ότι όλοι μας είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε για να έχουμε κοινή αξιολόγηση κινδύνου για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να γίνει υπό την αιγύδα της Γενικής Διεύθυνσης HOME. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων αυτών ε, που είναι ε, τα πιο πλούσια όσον αφορά τις ε, στρατιωτικές πληροφορίες, συμφώνησαν να συνεργαστούν υπό την αιγύδα της Γενικής Διεύθυνσης HOME, ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή αξιολόγηση κινδύνου για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμφωνήσαμε το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης κινδύνου να δημοσιευτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας ε, της Αεροπορίας. Θα διαβιβαστεί σε όλα τα κράτη-μέλη και στις ε, ε, αεροπορικές εταιρείες για να προειδοποιηθούν σχετικά με πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση υπέρπτυσης συγκεκριμένων περιοχών. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι αποτελεί ευθύνη των αεροπορικών εταιριών να λάβουν τις αποφάσεις τους με βάση αυτές τις πληροφορίες. Δηλαδή, το αν θα έχουν συγκεκριμένε διαδικασίε, το αν θα έχουν μέτρα μετριασμού του κινδύνου κλπ. Ε, αυτό αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό ήταν σημαντικό αποτέλεσμα τη ομάδα μα. Επίσης, ε, καθορίσαμε τους μηχανισμούς ε, για επίγουσε περιστάσει Σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχουμε το χρόνο να δημιουργήσουμε μια ε, ομάδα εργασίας ε, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Home, να υπάρξει γρήγορη διαβούλευση των κρατών μελών ε, μέσω του διαδικτύου και να εκδώσουμε επιγόντως να ανακοινωθέν το, από πλευρά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια τη Αεροπορία. Εγώ ήμουν πολύ ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα αυτό, διότι όταν ξεκινήσαμε τι συζητήσει, δεν ήταν αυτονόητο ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. όσον αφορά τις ευθύνες ε, των ε, διαφόρων παραγόντων. Συστήνουμε σε κάθε κράτος μέλος ε, να δημιουργήσει εθνικό σύστημα αξιολόγησης κινδύνου. Όποτε λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις απειλές, θα πρέπει αυτές τις πληροφορίες να τις επεξεργαστούν οι κυβερνητικές ε, αρχές ε, και να συζητηθούν και με τις αεροπορικές γραμμές. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μοιράζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν ε, από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους με άλλα κράτη-μέλη και όποτε υπάρχει επίγουσα περίσταση θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμεύονται να κινηθούν γρήγορα με βάση τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Αεροπορίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη να ε, δημιουργήσει ε, σχέδιο υπό την ε, αιγύδα της Γενικής Διευθυνσής HOME και οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν την ευθύνη να υποβάλουν στις εθνικές αρχές, στην ΕΑΣΑ ή στο δίκτυο τους πληροφορίες που έχουν, αλλά εναπόκειται στις αεροπορικές εταιρείες να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το τι θα κάνουν. Επίσης, η ΕΑΣΑ δημοσιεύει πληροφορίες και συστάσεις με βάση την κοινή αξιολόγηση κινδύνου. Και επίσης, θα υπάρχει ο μηχανισμός ε, για επίγουσες ε, περιστάσεις. Αυτή λοιπόν η ειδική ομάδα ε, είχε εκπροσώπου από κάποια κρατημέλη, όχι όμω και από το 28. Τώρα θα πρέπει να συντονίσουμε τι δράσει μα. Το σχέδιο μα είναι να παρουσιάσουμε τις συστάσεις μας ε, στη, στο Διευθυντικό Συμβούλιο μας ε, τον Ιούνιο, όπου εκπροσωπούνται και τα 28 κράτη-μέλη και μόλις έχουμε το πράσινο φως να ξεκινήσουμε να ε, εφαρμόζουμε το σχέδιο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε νέα υποδομή, θα πρέπει να γίνουν κάποιες δοκιμές, να δημιουργηθεί το δίκτυο για το οποίο μιλάμε Νομίζω όμως ότι όλα αυτά ε, είναι πολύ φυσιολογικά. Επίσης, ε, έχουμε ε, το δελτίο μας για τη διαβίβαση πληροφοριών. Πιστεύουμε ότι λειτουργεί καλά και επίσης εξετάζουμε την δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης αντίδρασης για να μπορούμε να απαντούμε σε αιτήματα 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω τη δική σας υποστήριξη για ε, κάτι. Αναθεωρούμε τον βασικό κανονισμό, όπως ανέφερα και πριν. Και ως αποτέλεσμα έχουμε εισάγει ένα συγκεκριμένο άρθρο το οποίο ε, αφορά το μηχανισμό αυτόν και ελπίζω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσά ώστε να λειτουργήσει αυτό τελικά διότι όπως πάντα μερικές φορές είναι δύσκολο να περάσει από το Συμβούλιο κάτι που έχουμε συμφωνήσει στην ειδική ομάδα. Κάποια κράτη-μέλη λοιπόν ε, συμφώνησαν στην ειδική ομάδα, αλλά ε, στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου φαίνεται να διστάζουν. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε να μα στηρίξετε. Πρόκειται για συλλογική προσπάθεια. Και προσβλέπω στην υποστήριξή σας, διότι είναι ένα θέμα στο οποίο ε, πρέπει αναγκαστικά να ε, ενεργήσουμε ως Ευρωπαίοι και να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο για να ε, μειώσουμε τον κίνδυνο για την αεροπλοεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κύη για αυτή την παρουσίαση και φυσικά θα έχετε την υποστήριξή μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή λύση σε αυτό τουλάχιστον το θέμα. Είπατε ότι θα ασχοληθεί με αυτό η DG Home. Πού είναι η DG Home? Είναι η Γενική Διεύθυνση του Επιτρόπου για Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις. Ο οποίος ε, επίτροπος είναι ο κύριος Αβραμόπουλος. Και ο Γενικός ε, Διευθυντής είναι ο Ματίας Ρούιτε, πολύ γνωστός, που ήταν στη γραμματεία της Επιτροπής μας. Ο κύριος Βίν Φαντεκάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνετε ότι ως Ολλανδός Ευρωβουλευτής ενδιαφέρομαι πάρα πολύ ε, για τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας ε, το 2015 είπε κατά λάθο ο κύριος ε, Κί και αυτό είναι ενδεικτικό γιατί ήταν τον Ιούλιο του 2014 και δείχνει προσοχή, έχει σημασία αυτό διότι τα θύματα και οι οικογένειες δηλαδή και οι δικοί τους είναι πάρα πολύ ανυπόμονοι. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, έρευνες ε, και ακόμα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τα δεδομένα των ραντάρ από τη Ρωσία, την Ουκρανία και πάει λέγοντας. Και γνωρίζω ότι τώρα δεν μπορείτε να πείτε ίσως κάτι γι' αυτά, αλλά σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που μπορεί να καθησυχάσει ή να μετριάσει λίγο την ανυπομονησία των συγγενών, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Είναι καλό αυτό που μας παρουσιάσατε, ωραία, ότι η Task Force έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά στην ουσία, περί τίνος πρόκειται, όπως και σε πολλά ευρωπαϊκά εγχειρήματα, θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμόζονται και να έχουν και αποτελέσματα. Εγώ έχω μια ερώτηση για τις αρμοδιότητες της ΕΑΣΑ. Ο κύριος Κι λέει, προσοχή, ο κύριος Μαρινέσκου στην έκθεσή του να δώσει προσοχή ε, στις δικές σας επιθυμίες και τα μελήματα που μας παρουσιάσετε συμπεράσματα. Έχω όμως την εξή ερώτηση. Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Αυτά όλα που ζητάτε έχουν οικονομικές συνέπειες, χρειάζονται περισσότερο προλογισμό αρκεί ο, ο Έχω την αίσθηση ότι η ΆΣΑ έχει ένα σωρό καθήκοντα που πρέπει να καλύψει με τον υφιστάμενο προπολογισμό και πρέπει να το μελετήσουμε αυτό. Μετά, Πρόεδρε, η Γενική Διεύθυνση Χώου μεσωτερικών για ποιο λόγο να επιληφθεί. Γιατί όχι η DG Move που είναι για τις μεταφορές. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών ε, θα πρέπει να κάνει όλη τη βρωμοδουλειά, για να το πω έτσι, και μετά για τις αρμοδιότητες πηγαίνουν όλοι στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Νομίζω ότι δεν είναι καλή η κατανομή αρμοδιοτήτων. Αυτά σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ πάντως για τη δουλειά που κάνετε και για τη συνεργασία της ε, ομάδας δράσης και ελπίζω να μπορέσουμε έτσι να αποφύγουμε και νέες τραγωδίες. Ευχαριστώ πολύ. Ρόμπετ Ζήλα. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ αναλυτική παρουσίαση και την πρόταση που μας κάνατε. Αλλά για αυτά που υποβήμα για την ιδιαίτερη κατάσταση του MH17 διότι στα δυτικά μέσα ενημέρωσης Ορισμένοι ε, αναφέρουν, ορισμένοι μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν ήταν πύραυλος εδάφους αέρος, αλλά αέρος αέρος μετά την, ε, τις προσεκτικές δηλώσεις κάποιων από αυτούς που διερευνούν το επεισόδιο αυτό, όλα αυτά δημιουργούν μεγάλη σύγχυση. Αλλά για αυτή την ειδική ομάδα, δύο ερωτήσεις. Οι μεγαλύτερες χώρες ε, της Ένωσης που έχουν ε, υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν ε, να έχουν πληροφορίες αλλά ορισμένες φορές δεν λαμβάνουν τις ίδιες προφορίες ε, και δεν τις στέλνουν, δεν στέλνουν τις ίδιες προφορίες στα σύστημά σας. Ποιος τις αποτιμά και ποιος τελικά βγάζει ένα πόρισμα για να ενημερώσει περαιτέρω. Εντός της ε, EASA ποιος κάνει την αποτίμηση, την αξιολόγηση των πληροφοριών γιατί αν ε, οι αεροπορικές εταιρείες ε, λαμβάνουν ε, αντικρουόμενε προφορίες δεν μπορούν να αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη, ποια είναι η πιο αξιόπιστη. Επίση, περιγράψατε πώς προτίθεστε να ε, ανταλλάσσετε αυτή την πληροφόρηση με τα κράτη-μέλη και του εθνικού αερομεταφορεί. Τι πρόκειται να κάνετε με τις αεροπορικές εταιρείες των τρίτων κρατών. Γιατί ξέρετε αυτό αφορά του πολίτε μα, γιατί και οι πολίτε μα μπορεί να πάρουν την αεροφλότη, την μαλέζουν. Αυτές οι ερωτήσεις. Γκεζίνε Μάσινα. Ευχαριστώ. Από πλευρά των φιλελευθέρων, Κυριακή, σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μας στείλετε αυτή την παρουσίαση. Παρακαλώ να μας τη στείλετε. Ωραία. Ωραία, ήθελα να βεβαιωθώ. Και να αναφέρω για τις ε, τρίτες χώρες αυτό που είπε και ο Ρόμπερτ Ζήλε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά αυτά που επιτύχατε γιατί επιτύχατε να υποχρεώσετε να γίνεται ανταλλαγή ή μάλλον να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Σε άλλους τομείς όπως η καταπολέμηση τρομοκρατίας δεν το καταφέραμε. Ξέρετε η τρομοκρατία έχει πολλές εκφάνσεις και δεν ανταλλάσσουν τα κράτη-μέλη πληροφορίες Βεβαίως εμένα δεν μου αρέσει το PNR να συλλέγουμε τα στοιχεία όλων των πολιτών της Ένωσης και να ανταλλάσσουμε όλα τα στοιχεία. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εγκρίθηκε το PNR όπως εγκρίθηκε. Αλλά και σε αυτό το θέμα τα κράτη-μέλη ήταν κατά της ε, ε ανταλλαγής πολλών προφοριών. Αλλά, εν περιπτώσει, το βασικό μου ερώτημα είναι τι ρόλο θα παίξει από εδώ και μπρο το P1. Θα ξεκινήσετε τον ε, Ιούνιο την εφαρμογή. Είναι καλό που θα αρχίσει γρήγορη εφαρμογή. Και όταν θα εφαρμοστεί πλήρω το PNR, θα παίξει ρόλο στι προσπάθειέ σα ή χρειάζεστε πολύ διαφορετικέ προφορίε για του πραγματικού κινδύνου στι εμπόλεμε περιοχέ ή για συγκεκριμένα άτομα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η Μαρία Κίλεν. Κίλανεν. Ευχαριστώ πολύ για τη σημαντική ενημέρωση που μόλις λάβαμε. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Μάισνερ. Πού έχετε τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, τις περισσότερες δυσχέρειες. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία να είναι κατηγορηματικά κατά της πλήρους ανταλλαγής προφοριών και που κάνουν ό,τι μπορούν για να την παρεμποδίσουν. Θα θέλαμε να το μάθουμε αυτό, ούτω ώστε να ξέρουμε ποιους εμείς πρέπει να πιέσουμε. Ούτω ώστε αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών να γίνει ουσιαστικό μέσο. Αυτό είναι αναγκαίο, οπωσδήποτε. Ούτω ώστε να μην προκύψει μια κατάσταση όπου όλοι μας οι πολίτες θα θεωρούνται ύποπτοι τρομοκρατίας ούτως ώστε όλοι να αισθάνονται ότι τους αντιμετωπίζουν ως υπόπτους ε, στις, ε, στους ελέγχους. Η Καρίν Μεντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και κύριε Κύ για την παρουσίασή σας. Διαβάζοντας την έκθεσή σας, συμφωνώ που λέτε ότι το καλύτερο επίπεδο για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά το ότι κάθε κράτος μέλος θα κάνει τις δικές του αξιολογήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Γιατί έχω την εντύπωση ότι προσθέτουμε ένα επιπλέον επίπεδο, μία επιπλέον φάση συντονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση κρίσης, όταν πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα, θεωρούμε ότι θα είναι αποτελεσματική αυτή η διαδικασία. Γιατί η ΕΑΣΑ δεν θα μπορούσε ε, να παίξει εκείνη το ρόλο του συντονιστή αντί για την Κομισιόν. Η ΕΑΣΑ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι σε θέση να συλλέξει σύντομα τις προφορίες από εμπόλεμες περιοχές, όταν προκυπτούν κίνδυνοι με την υπερπτήση κάποιας περιοχής. Μήπως για αυτή ακριβώς τη φάση, κύριε εκεί, θα μπορούσατε να μου δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πέτε ε, που είναι και ο τελευταίος συντονιστή, ε, πριν περάσουμε μετά σε όσους συναδέλφου έχουν ζητήσει το λόγο. Αλλά πριν από όλα αυτά, να ε, καλωσορίσω μία ομάδα επισκεπτών από το Πανεπιστήμιο του Βισμπάντεν, τη Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών, που την έχει προσκαλέσει ο κύριος Μίχαελ Γκάλαρ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ η κυρία Φώστερ και ευχαριστώ και τον κύριο Κι για την παρουσία του. Ορισμένες λοιπόν παρατηρήσεις. Όλοι προσπαθούμε να αντιδράσουμε τάχιστα μετά από αυτή την τρομοκρατική επίθεση γιατί δεν ήταν ε, αεροπορικό ατύχημα ήταν ε, η θελημένη τρομοκρατική απόπειρα. Ε, αν τώρα κατάλαβαν περί τι αεροσκάφους και τι εταιρεία σε πρόκειτο, αυτό είναι άλλο θέμα έχω τις εξής ανησυχίες. Αναφέρατε ποια γενική διεύθυνση θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Η DigiMove και η DigiTran έχουν αντιμετωπίσει τα θέματα ασφάλειας στα αεροδρόμια. Όσο ε, άρχιζε να λειτουργεί η ΕΑΣΑ τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνω όμως γιατί αναφέρεται και την DG Home αλλά δεν επικρίνω εσάς, αλλά αυτά που ε, ακούστηκαν. Γιατί νομίζω ότι εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και αν θέλουμε να αντιδράσουμε σύντομα, πώς θα αντιδράσουμε σύντομα. Όταν διάφορες υπηρεσίες, φορείς, οργανισμοί πρέπει να κάνουν διάφορα πράγματα. Μας ενδιαφέρει ταχύτητα αντίδρασης. Όταν κάνουμε αξιολόγηση των κινδύνων, Βέβαια μπορούν να ασχοληθούν πολλές υπηρεσίες. Αλλά η αντιμετώπιση μας πρέπει να βασίζεται ακριβώς πάντα στην αντιμετώπιση του κινδύνου. Και μετά ο αερομεταφορέας θα πάρει την απόφαση. Και αυτές τις αποφάσεις μπορεί να τις πάρει μόνο με βάση την πληροφόρηση που θα έχει λάβει από τα κράτη-μέλη. Όπως είπατε όμως, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που ε, διατρέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από άλλα για μια σειρά από ιστορικούς ή συγκυριακούς λόγους. Και όλοι συμφωνούμε. Θα πάμε να επισκεφθούμε τον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας σε δύο εβδομάδες και θα το συζητήσουμε και με εκείνους. Αλλά είναι λίγο κατακαιρματισμένες οι προσπάθειές μας. Δηλαδή ορισμένοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, άλλοι λένε πρέπει να κάνουμε το άλλο. Το θέμα όμως είναι ότι ακόμη και αν είχαμε όλα αυτά τα μέτρα, δεν νομίζω ότι θα είχαμε αποτρέψει αυτή την επίθεση. Γιατί άμα υπάρχουν τέτοιοι που παίζουν τέτοιο ρόλο, που είναι ανεξέλεγκτοι όπω η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μπορεί να κάνουν εκτοξεύσεις δοκιμών, πυράβλων. Άρα το βασικό είναι οι υπηρεσίες καταπολέμησης τρομοκρατία να έχουν την αναγκαία ενημέρωση και να μπορούν να την ανταλλάξουν. Και κάποιοι διστάζουν πιστεύω. Ορισμένοι από αυτούς που θα έπρεπε να παίξουν κύριο ρόλο. Γιατί φοβούνται ότι αν ανταλλάξουν πληροφορίες, οι πληροφορίες αυτές δεν θα μείνουν απόρριτες. Εδώ υπάρχουν κάποια θέματα πιστεύω. Και καταλήγοντας, σωστό είναι αυτό που υπόθηκε για την ε, χρηματοδότηση, τον προϋπολογισμό της ΕΑΣΑ. Ξέρουμε ότι τα τρία τέταρτα του οργανισμού της χρηματοδότησής σας ε, προκύπτουν από τον ε, κλάδο τον ίδιο. Ενώ εμείς συμβάλλουμε λίγο σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να κάνουμε πιο μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ΕΑΣΑ. Εφόσον θέλουμε η ΕΑΣΑ να κάνει τόσο περισσότερα για να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, δεν μπορούμε να τα κάνουμε πενταροδεκάρες. Ξέρετε ότι μπορεί να έχω επικρίνει για άλλα θέματα την ΕΑΣΑ, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει πολύ πιο σίγουρη χρηματοδότηση. Γιατί αναφερθήκατε και στα ανεπάδροτα αεροσκάφη, τα drone. Και όσον αφορά τον κανονισμό για την ΕΑΣΑ, για τον οποίο είμαι σκιώδης εγώ από πλευράς της ομάδας μου, της ECR, και θέλουμε να το δούμε λεπτομεριακά, μπορούμε να το συζητήσουμε και μεταξύ μας. Αλλά στα πλαίσια των περιορισμών ε, που έχετε, έχετε κάνει πολλά πιστεύω, αρκετά σύντομα, αλλά ανησυχώ γιατί υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φορείς, η μία γενική διεύθυνση, ο άλλος φορέας. Μα πόσο δεν πλακούν σε κάθε απόφαση. Με ανησυχεί πολύ αυτό. Και πιστεύω ότι πρέπει να επιχειρούμε να προλαμβάνουμε και όχι να αντιδρούμε. Άρα οι διαδικασίες μου φαίνονται υπερβολικά βαριές. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πάντα με τις διαδικασίες της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι λάβατε υπόψη τις συστάσεις που κάναμε όταν το πρώτο συζητήσαμε μετά από αυτή την τρομοκρατική επίθεση και πιστεύω ότι όλοι θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Λου, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κι για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες της Ευρώπης να έχουμε συντονισμένη ε, απάντηση σε αυτή την επίθεση, γιατί τώρα είναι δύσκολη καιρή ε, ε, από τότε που έγινε αυτή η επίθεση έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και θα πρέπει και οι επιβάτες και οι πολίτες γενικότερα να γνωρίζουν ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους προστατεύουμε. Πολλές ανησυχίες εξέφρασαν ε, συνάδελφοι και συμμερίζομαι για τα κράτη-μέλη, για τις μυστικές υπηρεσίες, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Πρόσφατες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις της Βρυξέλλης και το Παρίσι το κατέδειξαν αυτό. Εδώ δεν ε, θέλω να στιγματίσω οποιαδήποτε χώρα, αλλά όταν έχουμε 28 κράτη-μέλη, καταλαβαίνετε ότι ο καθένας δεν έχει την ίδια ε, δυνατότητα μυστικών υπηρεσιών ε, και του στρατού και των υπολείπων υπηρεσιών, ούτε την ίδια δυνατότητα απόκρισης. Αυτό μπορεί να είναι εμπόδιο λοιπόν. Δεν ξέρω, το έχετε αντιμετωπίσει, δεν το έχετε αντιμετωπίσει, έχετε πλήρη πρόσβαση, δεν έχετε στις πληροφορίε αυτές. Είναι ανησυχία ειλικρινής δική μας, θα μπορούσατε να μας απαντήσετε. Ε, αναφερθήκατε λίγο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό εννοούσατε. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανταλλάσσονται πληροφορίε. Μιλήσατε και για τι αεροπορικέ εταιρείε που θα πρέπει να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα μέσα σε ώρε, ημέρε. Όταν τίθεται ένα ζήτημα επίθεση ε, ή προειδοποίηση, σύμφωνα με τη δική σα εμπειρία, έχουν αυτή τη δυνατότητα οι εταιρείε να αντιδρούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ενώ το προσωπικό, τους πόρους, ε, τις δυνατότητες πληροφόρησης. Αναγνωρίζω ότι αυτό θα σημάνει περισσότερο φόρτο εργασίας ε, για το δικό σας οργανισμό και θα χρειαστεί ενδεχομένως και μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Γιατί σας ζητούμε να κάνετε περισσότερα στην ασφάλεια των επιβατών, είτε αυτό είναι ε, πτήση στα αεροδρόμια, η ασφάλεια των ελέγχων κτλ. Γίνεται αυτό με τους υφιστάμενους οικονομικούς πόρους. Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Χρειάζεστε άλλη υποστήριξη από πλευράς μας. Θα σας υποστηρίξουμε όσο μπορούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ο Ματίας Φαν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κι για την ε, ξεκάθαρη παρουσίασή του. Είναι σαφές, το άκουσε και ο Βίμ Φάντεγκα, τον ανέφερε, ότι έχουν περάσει τόσοι μήνες και δεν υπάρχει σύστημα ευρωπαϊκής προειδοποίησης. Ε, μας λέτε ότι θα γίνει. Πότε. Έχω ερωτήσεις. Πρώτον, όταν δίνετε συμβουλές και οδηγίες στις αεροπορικές εταιρείες, αυτό είναι απολύτως εθελοντικό. Είναι στη διακριτική τους ευχαίρεια. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε ένα δεσμευτικό χαρακτήρα σε αυτές τις συμβουλές ποιος έχει το τελευταίο λόγο. Υπηρεσίες ε, πολιτικής αεροπορίας των κρατών μελών ε, μπορούν ε, να απαγορεύσουν σε κάποιες αεροπορικές εταιρείες να περάσουν από μια συγκεκριμένη διαδρομή ή ας ΑΣΑ θα το κάνει αυτό. Ποιος το αναλαμβάνει. Και γίνεται μια πρόταση για να θεώρηση του βασικού κανονισμού του οργανισμού σας αν θέλουμε εμείς να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης, δεν πρέπει να το αναφέρει αυτός ο κανονισμός ότι οι δικές σας οδηγίες θα πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Χρειάζεται δηλαδή να γίνει πιο αυστηρή η πρόταση και πώς θα έχει διατύπωση. Αυτά προς το παρόν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια ερώτηση έχω προς τον κύριο Κίκη και μόνο. Στις κάτω χώρες και σε άλλες χώρες ζουν εκατοντάδες συγγενείς των θυμάτων. Και υπάρχει σύστημα που θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την τραγωδία. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε στους συγγενείς ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί τέτοια τραγωδία. Εκατοντάδες ήταν οι νεκροί. Περί αυτού πρόκειται. Θα έχουμε ένα σύστημα τώρα που στα χαρτιά θα είναι τέλειο και φανταστικό. Είναι όμως αυτό το σύστημα που μπορούμε να πούμε στα θύματα και στους συγγενείς και να τους διαβεβαιώσουμε ότι αποκλείεται Ε, ε, πλέον ε, οι τρομοκράτες στην Ανατολική Ουκρανία να ξαναεκτοξεύσουν πύραυλο μπουκ κατά αντίστοιχου αεροσκάφους. Η απάντηση είναι όχι. Πρόεδρε, εδώ και χρόνια τα ξέρω αυτά, γιατί έχω δουλέψει στην επιθεώρηση της πολιτικής αεροπορίας της κάτω χώρας. Και ξέρουμε ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν δίνουν τις πληροφορίες στην πολιτική αεροπορία. Ξέρουμε και το έχουμε ζήσει ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι ίδιες. Άλλοι οι Αγγλικοί, άλλοι οι Βουλγαρικοί ας πούμε, ένα παράδειγμα σας αναφέρω. Και έχουμε εμπειρία ε, ότι εντάξει αυτή η εταιρεία ήταν μη κοινοτική. Μπορεί να ήταν κοινή πτήση με την KLM ε, της Μαλέσιαν, αλλά δεν ήταν ο αερομεταφορέας ευρωπαϊκός. Δεν ήταν αυτό που λέμε EU carrier. Τώρα θα επέλθει η λύτρωση από αυτά που μας ε, συνιστάτε. Δεν νομίζω. Είναι πάρα πολύ ωραία στα χαρτιά, αλλά δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Ούτε πρόκειται να αποτρέψει νέα τραγωδία. Δεν το πιστεύω καθόλου ότι αυτό το σύστημα είναι λύση. Και δεν πρόκειται να είναι λύση, διότι εδώ μιλάμε για μυστικές υπηρεσίες που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, που εργάζονται διαφορετικά και δίνουν ψήγματα ε, πληροφορίας ε, μοιράζονται. Και μάλιστα τα δίνουν μόνο με αντάλλαγμα. Θα σου πω κάτι να μου πεις και εσύ όμως. Έχω πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορούμε να αποτρέψουμε στο μέλλον τέτοιου είδους τραγωδίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Ε, σας δίνω το λόγο και μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς καταλήξατε στην απόφαση ε, να γίνουν όλα υπό την αιγίδα της ε, Γενικής Διεύθυνσης Home. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Ε, καταρχάς, ε, ζητώ συγγνώμη, είναι πράγματι το ατύχημα συνέβη το 2014. Μπερδεύτηκα. θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει το ατύχημα. Αυτό αναρωτιόμαστε κάθε φορά που ε, έχουμε ένα ατύχημα. Το ίδιο στην περίπτωση του ατυχήματος ε, του αεροπλάνου της German Wings. Είναι αδύνατο να πει κανείς ότι κάτι τέτοιο δεν θα ε, ξανασυμβεί ποτέ. Αλλά για να σας δείξω πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι λειτουργούν σήμερα άτυπα και με βάση την καλή βούληση διαφόρων να μοιραστούν τις πληροφορίες που έχουν, αλλά λειτουργεί το σύστημα. Τι συμβαίνει λοιπόν. Μία χώρα λέει ότι έχουμε ενδείξεις για μια ε, τρομοκρατική ομάδα που με τα συγκεκριμένα όπλα η οποία μετακινείται προς μια περιοχή. και αυτό μπορεί να επηρεάζει την κίνηση γύρω από ένα αεροδρόμιο ή μια συγκεκριμένη περιοχή. Διότι ξέρουμε ότι τα συγκεκριμένα όπλα έχουν ε, συγκεκριμένο βεληνικές. Αλλά παλαιότερα τις πληροφορίες αυτές τις είχε ένα ε, κράτος μέλος, ενώ τώρα πια μοιραζόμαστε τις πληροφορίες αυτές και το σύστημα λειτουργεί. Αποτρέπουμε ατυχήματα. Δεν το ξέρουμε αυτό, διότι δεν συμβαίνουν. παρέχουμε καλύτερες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο κινδύνου στις αεροπορικές εταιρείες. Από ό,τι γνωρίζουμε, ναι. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν θα ξανασυμβεί τέτοιο ατύχημα στο μέλλον. Αλλά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να διαβιβάζουμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας ε, στους ε, αρμόδιους παράγοντες. Όσον αφορά τις ε, αεροπορικές εταιρείες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουμε τις πληροφορίες αυτές στις ε, αεροπορικές εταιρείες Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς φορείς όπως είναι η ΆΤΑ. Επίσης, συνομιλούμε με άλλα κράτη για να δούμε αν θέλουν ε, να έχουν ανταλλαγή πληροφοριών μαζί μας, ε, αν θέλουν να μας δώσουν εκείνες πληροφορίες ή να έχουν πρόσβαση στις δικές μας. Εργαζόμαστε πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης, συνομιλούμε με τους αερομεταφορείς, ώστε εάν θεωρήσουν ότι υπάρχει κίνδυνος, να είναι υποχρεωτικό, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, να έχουν την ευθύνη να μοιραστούν τις πληροφορίες με τους εταίρους τους. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε όσο γίνεται ευρύτερο κύκλο ανθρώπων Και φυσικά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, ε, αεροπορικές εταιρείες εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιβάτες πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αγοράσει εισιτήριο με ευρωπαϊκή εταιρεία. Όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, χρειάζεται ένα ασφαλές δίκαιο, χρειάζονται ειδικοί χώροι, πρέπει να καλύψει κανείς όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρώπης και η Γενική Διεύθυνση MOVE δεν έχει πρόσβαση σε όλα αυτά. Ε, τέτοια πρόσβαση έχει η Γενική Διεύθυνση HOME. Συνεργαζόμαστε στενά λοιπόν με τη Γενική Διεύθυνση αυτή. Όπως ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, ο ματία Ρίτερ γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα μεταφορών. Ε, έχουμε πολύ καλή σχέση και λειτουργεί καλά η συνεργασία. Μία από τις δυσκολίες που αναφέρατε κιόλας είναι ότι η ομάδα της DG Home ε, έχει συνάντηση τέσσερις φορές το χρόνο. Ή ε, κατόπιν συγκεκριμένης αφορμής, όπως ε, για παράδειγμα την τρομοκρατική επίθεση στο αεροσκάφος της Metrojet στην Αίγυπτο. Απαιτείται όμως κάποιος χρόνος να οργανωθούν οι συναντήσεις αυτές και να έρθουν όλες στις Βρυξέλλες ή να οργανώσουμε ε, ασφαλή τηλεδιάσκεψη. Κατά τις ε, συναντήσεις της ομάδας αυτής εξετάζουμε τα συστημικά προβλήματα. Ποια είναι η κατάσταση στην Αίγυπτο, στο Πακιστάν, στο Ιράν, το Ιράκ κλπ τι εξελίξεις έχουμε, τι κίνδυνος βλέπουμε να υπάρχει στα αεροδρόμια, στον εναέριο χώρο. Και με βάση τις πληροφορίες μας, διαμορφώνουμε την κοινή θέση που δημοσιεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Αεροπορίας. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, δεν λαμβάνει η όλες τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη ε, και τις αναλύει τα κράτη-μέλη όλα μαζί στην ομάδα εργασίας αυτή καταλήγουν σε κοινή θέση όσον αφορά τον κίνδυνο. Στην ειδική ομάδα είχαμε συζήτηση σχετικά με το τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν έχουμε ε, κοινή γνώμη όσον αφορά τον κίνδυνο. Σε τέτοια περίπτωση θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά ε, εντός ε, του ΕΑΣΑ θέλουμε να δημοσιεύουμε τις πληροφορίες που έχουμε με τις διαφορετικές θέσεις που υπάρχουν, ώστε οι αερομεταφορείς να έχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια και Αεροπορία δεν είναι ο οργανισμό μυστικών πληροφοριών, παρότι έχουμε προσωπικό με τέτοιε δυνατότητε. Βασιζόμαστε στα κράτη-μέλη ε, και στην ε, κοινή ε, αξιολόγηση κινδύνου στην οποία καταλήγουν. Αυτό μπορεί να μην είναι αρκετά προορατικό σε περίπτωση επίγουσας κατάστασης και τους προηγούμενους μήνες είδαμε πυράβλους στην Κασπία προς την Συρία. Είδαμε δοκιμές βαλιστικών πυράβλων στο Ιράν Είδαμε περιπτώσεις όπου έπρεπε να αντιδράσουμε εντός ορών. Σε τέτοιες περιπτώσεις ε, δεν έχουμε την δυνατότητα να περάσουμε την κανονική διαδικασία μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Home. Αλλά μέχρι τώρα αυτό που κάναμε ήταν ότι ε, έχουμε ένα δίκτυο επαφών σε όλα τα κράτη-μέλη και θέτουμε την ερώτηση. Λάβαμε αυτές τις πληροφορίες, ε, ποια είναι η θέση σας, τι πρέπει να κάνουμε. Και φυσικά προτείνουμε διάφορες λύσεις. Αυτό έχει λειτουργήσει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Και στις δύο περιπτώσεις ο ΕΑΣΑ μπόρεσε να εκδώσει σύσταση εντός ορών. Λειτουργεί λοιπόν το σύστημα. Μία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν ε, πρέπει να εκδίδουμε συστάσεις. Ε, ή υποχρεωτικές ε, εντολές. Ε, δεν ε, υπάρχει δυνατότητα ο οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει στο έδαφος τα αεροσκάφη. Αν και αυτό γίνεται στην περίπτωση της Airbus. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη το να πει κανεί ότι δεν θα υπάρξουν πτήσεις προς την περιοχή αυτή. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα αυτή συχνά. Δεν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, τη δυνατότητα αυτή, ωστόσο προτάθηκε στο κείμενο που θα δείτε, την αναθεώρηση του βασικού κανονισμού δηλαδή, διότι σε κάποια κράτη-μέλη είναι ο μόνος τρόπος να εμποδίσουμε τους αερομεταφορείς να έχουν πτήσεις προς κάποια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου για παράδειγμα στις κάτω χώρες. Η Ολλανδική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει την πολιτική αρμοδιότητα να απαγορεύσει σε κάποιον αερομεταφορέα υπερπτήσει συγκεκριμένες περιοχές. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, στη Γαλλία, στην ε, Γερμανία, όχι όμω ε, στι κατοχώρε, στι σκανδιναβικέ χώρε, Βουλγαρία κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα ε, τι κοινέ ανάγκε ε, όλων των ε, παραγόντων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται ακριβώ να θέσουμε αυτό το θέμα τη ευθύνη. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να βασίζεται σε ευρεία διαβούλευση με όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να συμφωνούν τα κράτη-μέλη μεταξύ του. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε στην πράξη. θέσατε κάποιες ερωτήσεις ε, σχετικά με το ατύχημα που αφορά την πτήση ε, MH17. Ε, δεν ερευνήσαμε εμείς το συγκεκριμένο ατύχημα. Υπάρχει η ομάδα των κάτω χωρών που διαρευνεί το ατύχημα. Έκανα μια δήλωση στο Κοινοβούλιο των κάτω χωρών πριν κάποιους μήνες. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Δεν έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Όσον αφορά τους πόρους μας, και το αν συμπεριλαμβάνεται στην εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και της Αεροπορίας ε, να ε, ασχολείται με τέτοια θέματα. Είχαμε κάποιες ε, θεωρητικές συζητήσεις με κάποια κράτη-μέλη. Μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε κάτι τέτοιο, διότι η εντολή σας δεν συμπεριλαμβάνει θέματα ασφαλείας. Νομίζω ότι ήδη το ανέφερα στην Επιτροπή σας. Το θέμα είναι ότι η υπέρπτυση κάποιες περιοχής έχει να κάνει με την ασφάλεια των επιβατών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναλαμβάνουμε δράση για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Η απάντησή μου λοιπόν ήταν, παρότι μπορεί, ε, εάν δει κανεί αυστηρά την εντολή μα, να μην ε, συμπεριλαμβάνεται στην εντολή μα, ε, έχει να κάνει με την ασφάλεια των επιβατών στην πτήση. Ε, και άλλωστε, εάν δεν το κάνει αυτό ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Αεροπορία, ποιο θα το κάνει, η Γενική Διεύθυνση Home, η Γενική Διεύθυνση MOVE. Έχουμε τα εργαλεία για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα το κάνουν αυτό οι εθνικοί ε, φορεί. Φυσικά μπορούν να το κάνουν, αλλά όπως είπα νωρίτερα αυτό δεν αρκεί και δεν καλύπτει ε, το σύνολο των ε, Ευρωπαίων. Όσον αφορά τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε ε, προσωπικό στο οποίο βασιζόμαστε Προς το παρόν δεν έχουμε τόσο πολλές κρίσεις, περίπου μία κάθε τρίμηνο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προσλάβουμε ε, ομάδες ε, που να είναι διαθέσιμες 24 ώρε την εβδομάδα. 24 ε, ώρες το 24ωρο, συγγνώμη. Έχουμε όμως προσωπικό, διασφαλίζουμε την εύκολη πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, για παράδειγμα. Εάν όμως ε, αυξηθεί ο όγκος ε, δουλειάς μας, ε, κάτι που απέφχομαι, τότε μπορεί να χρειαστεί να έχουμε ομάδες που να είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, αλλά κάτι τέτοιο είναι πολύ δαπανηρό όσον αφορά το δυναμικό. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να έχουμε κάποιο αποθεματικό για να διατηρήσουμε ε, το επίπεδο του προσωπικού που έχουμε, αλλά δεν ζητάμε αύξηση του προϋπολογισμού, γιατί μπορούμε να καλύψουμε ε, τα καθήκοντά μας με ε, το προσωπικό που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τον ΙΚΑΟ, το σύστημα έχει ως εξής. Κάθε κράτος που ε, έχει αναλάβει δράση που αφορά κάποιο άλλο κράτο μέλο θα πρέπει να το δημοσιεύει. Για παράδειγμα, εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, αποφασίσουν ότι οι ε, αερομεταφορεί του δεν θα κάνουν υπερτήσει στη Συρία, θα πρέπει αυτό να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Και η Συρία έχει δικαίωμα να υποβάλει βέτο. Κάτι που περιορίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματο, αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα. Εμεί θέλαμε να είμαστε πιο προορατικοί, διότι αυτό το σύστημα ουσιαστικά είναι σύστημα αντίδραση. Δηλαδή, δημοσιεύεται μια απόφαση που έχει λάβει ένα κράτος, ε, ενώ εμείς θέλουμε να αξιολογείται ο κίνδυνος ε, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κίφ και για την παρουσίαση και για τις απαντήσεις σας. Ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα σας δούμε να μην είναι γιατί έχει προκύψει πάλι κάποια τραγωδία. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και παραλαμβάνω, ελπίζω να τα ξαναπούμε, αλλά όχι επειδή θα έχει προκύψει άλλη τραγωδία. Ο κύριος Φαντάλης. Πρόεδρε, μια ερώτηση στον κύριο Κι. Μίλησε για την έκθεση που πρόσφατα ε, παρουσιάστηκε στην Επίτροπο. Είναι διαθέσιμη η έκθεση αυτή και για τα μέλη του της Επιτροπής, Yes, it is. Μάλιστα, λέει ο κύριος Ωραία, ο πρόεδρος. Ε, είναι στο site μας. Μπορείτε να, το, να τη βρείτε στο website μας. Και πάλι ευχαριστώ και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μέρης διάταξη και περνάμε στην παρουσίαση του εγγράφου εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση του θορύβου από τη μεταφορά μέσω σιδηροδρόμου αγαθών. Η παρουσίαση αυτή θα γίνει από τον Ολιβιέ Ονιντή, στον οποίο με το λόγο. Σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Είναι η σημασία του θέματος ε, που σας ε, έπεισε ότι πρέπει να είμαι εδώ στο βήμα, αλλά οπωσδήποτε θέλουμε να σας κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση για τους ε, σιδηροδρομικούς θορύβους. Αυτό το θέμα επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια και θέλαμε να υπάρξει πρόοδος. Τα τέλη του 2015 υπήρξε ένα έγγραφο εργασίας προσωπικού για να συμπεριλάβουμε όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Θα είμαι σύντομος. Νομίζω ότι σας στείλαμε και ορισμένα στοιχεία στη γραμματεία για να είναι σαφές τι θέλουμε να παρουσιάσουμε. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ο θόρυβος είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα δημόσιας υγείας. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε επιπλέον προσπάθειες στον σιδοδρομικό κλάδο γι' αυτό, γιατί ξέρουμε ότι επηρεάζει και προκαλεί προβλήματα υγείας ε, σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Ποικίλει βέβαια από το ένα κράτο στο άλλο η σημασία αυτού του προβλήματος, αλλά βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ανησυχίε εντός του πληθυσμού. Το έγγραφο λοιπόν αυτό κάνει μια επισκόπηση των ενεργειών στο παρελθόν και προτείνει μεθόδους και μέτρα για να συμπληρώσουμε την εργαλειοθήκη που έχουμε στη διάθεσή μας. Δύο ιδιαιτερότητες. Πρώτη, είναι η βραδία προσαρμογή των νέων ε, βαγονιών, ούτως ώστε να έχουμε σιωπηλούς ε, μηχανισμούς πέδησης, που είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί ο κίνδυνος. Γιατί όπως ξέρετε, ένα βαγόνι μπορεί να λειτουργήσει 40-50 χρόνια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 40-50 χρόνια. Άρα η αναθεώρηση, συγγνώμη, ο επανεξοπλισμός των βαγονιών ε, παίρνει πολύ καιρό. Τα προβλήματα είναι διαφορετικής φύσης στην Ένωση και δεν θέλουμε να υπάρξει περαιτέρω κατακαιρματισμός σε ένα κλάδο όπου ήδη υπάρχουν υπερβολικές ρυθμίσεις και υπερβολική φραγμή ιδιαίτερα τεχνικής φύσης. Κάναμε μια σοβαρή μελέτη αντικτύπου που είναι στη διάθεσή σας όπου ε, κάναμε δοκιμές για μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνδυάζουμε μια σειρά από μεθόδους. Μία είναι οι επιδοτήσεις που δίνουμε με το παλιό καθεστώς TNT, αλλά και τώρα και με το CEF και μέσω των περιφερειακών χρηματοδοτήσεων. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κλάδο, ούτω ώστε να υπάρξει επανεξοπλισμός των βαγονιών. Ε, το πρώτο τμήμα, 20 εκατομμυρίων, έχει δοθεί με μία προκήρυξη και άλλα 20 θα προκηρυχθούν για τον ίδιο σκοπό. Επιπλέον, θα είδατε ότι όταν τα κράτη-μέλη προωθούν εθνικά προγράμματα, τα εξετάζουμε από τις ε, αρχές ανταγωνισμού μας ε, με θετική αρχική προσέγγιση. Ήδη δύο χώρες έχουν λάβει εξαίρεση από τις αρχές ανταγωνισμού για να επιταχυνθεί ο επανεξοπλισμός των βαγονιών. Τρίτο στοιχείο. Προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα. Υπήρχαν κάποια κίνητρα στο Recast, το οποίο έχετε προωθήσει, Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτά τα μέτρα, να υπάρξει διαφοροποίηση των τελών πρόσβασης ε, στις συνδρομικές γραμμές για να ενθαρρύνουμε τη χρήση αθόρυβων βαγονιών. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να χρεώνουν περισσότερο για τα βαγόνια που δεν έχουν αυτούς τους αθορύβους μηχανισμούς πέδησης και άρα κάνουν περισσότερο θόρυβο ούτω ώστε και εδώ να υπάρχει ένα σαφές οικονομικό κίνητρο για τις εταιρείες να επιταχύνουν τον, τις αλλαγές στα βαγόνια. Μπορούμε βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε και τις ε, επίσημες προδιαγραφές για την διαλειτουργικότητα. Από το 2005 σταδιακά έχουμε ορίσει ότι όλα τα νέα βαγόνια θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το ανώτατο όριο θορύβου που έχουμε προκαθορίσει. Σε μερικές μέρες θα ψηφίσετε συγκεκριμένα αυτή τη βδομάδα το τέταρτο σοδρομικό πακέτο και μάλιστα τον τεχνικό πυλώνα του όπου αναφέρουμε ότι έχουμε δυνατότητα και για υποχρεωτικό επανεξοπλισμό όχι μόνο λοιπόν τα νέα βαγόνια θα έχουν τους αναγκαίους νέους μηχανισμούς, αλλά θα είμαστε σαφώς και σε θέση να υποχρεώσουμε τις αλλαγές και στα υπάρχοντα παλιά βαγόνια. Ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν με βάση και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπουν ήδη κάποιες χώρες, η Γερμανία και η Ολλανδία και ενδεχομένω και η Γαλλία και η Αυστρία να προσθεθούν μέσω δικών τους εθνικών σχεδίων ε, με σαφείς προθεσμίες. θεωρούμε ότι αν εγκριθούν τα μέτρα αυτά νωρίς του χρόνου, τότε μέχρι το 2022 ίσως θα σταματήσει να υπάρχει δυνατότητα να κυκλοφορούν τα θορυβόδη βαγόνια. Θα υπάρχει βέβαια μια δυνατότητα εξαιρέσεων υπορισμένες ορισμένε προϋποθέσεις, δηλαδή ορισμένα βαγόνια που δεν συμμορφούνται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιοχέ όπου είναι χαμηλή η πυκνότητα του πληθυσμού. Έτσι θα δίναμε λίγο περισσότερο χρόνο σε ορισμένε χώρες όπου δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα γιατί οι συνδρομικέ γραμμές ε, δεν περνάνε πολύ κοντά από αστικά κέντρα. Πιστεύω ότι με όλες αυτές ε, τις άμεσες και έμεσες κινήσεις και κίνητρα και με μια σαφή πολιτική για αλλαγές σε όλα τα βαγόνια θα έχουμε ένα αποφασιστικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο ούτω ώστε να κλείσει αυτό το θέμα που για πολλά χρόνια μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Το λόγο έχει τώρα ο Βιμ Βανεκάμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσοι ήθιστε, και όσο μας έχει συνηθίσει, ο κύριος Ανίλη μας έχει κάνει μια πολύ καλή παρουσίαση και πολύ σαφή. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες όμως. Τώρα εδώ τι γίνεται. Μας δίνεται ένα κείμενο πολύ ωραίο, ανυπόγραφο κατά τα άλλα. Κάποιος με ρώτησε ε, μήπως το έχει δώσει κανένα λόμπι. Τι κείμενο είναι αυτό, ποιανού είναι. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω εγώ. Καλή ερώτηση. Το μεγαλύτερο λόμπι των Βρυξελών είναι αυτό, λέει ο κύριος Βαντάλεν και ο πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Ε, και η πίεση του Κοινοβουλίου θα σας βοηθήσει να το δημοσιεύσετε. Υποθέτω ότι σε όλες τις ιστοσελίδες της ε, Γενικής Διεύθυνσης MOVE θα δημοσιευτεί αυτό ως το πρόγραμμα δράσης, κύριε Ονίλη. Γιατί μας έχει πάρει τόσο χρόνο αυτή η ιστορία. Αυτή είναι η βασική ερώτηση και η κεντρική ιδέα. Ε, ε, μια ζωή ακούμε και από τον πρόεδρο να μιλάει για ποδήλατα και για το θόρυβο που κάνουν τα τρένα. Και είναι και το αγαπημένο του θέμα αυτό το θορύβο. Ε, μπορείτε λοιπόν να μου διασκεδάσετε αυτές τις αμφιβολίες. Δεύτερη ερώτηση. 20 εκατομμύρια στην πρώτη σεύκο, συν 20 ε, αργότερα, αν κατάλαβα καλά, σύνολο 40. Σωστά το κατάλαβα. Και τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η σχέση τώρα μεταξύ του τροχαίου υλικού, των βαγονιών, εν πάση περιπτώσει, ε, που μεταφέρουν εμπορεύματα και της υποδομής. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αν αλλάξουμε τις υποδομές, τις ράγες δηλαδή, μπορεί να μειωθεί ο θόρυβος καλύτερα και πιο γρήγορα και περισσότερο από ό,τι να περιμένουμε να αλλάξουν όλα τα βαγόνια. Και έχω και τέταρτη ερώτηση. Λέτε θα γίνει ε, και έρευνα. Συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό ε, Οργανισμό Σιδηροδρόμων και να ζητήσει μια δράση Ερευνητική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι είναι αυτό, ποιος θα το κάνει και πότε και ποια έρευνα είναι αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Πέτερ Βαντάλεν. Ευχαριστώ τον κύριο Νίλ για την παρουσίασή του. Το πρόβλημα με το σιδηρόδρομο είναι ότι έχουμε τριβή χάλιβα σε χάλιβα ε, και παράγονται πολλά δεσιμπέλ, αλλά και να μειωθούν πάλι θόρυβο θα κάνει ο χάλιβας που τρίβεται σε χάλιβα. Ε, καταλαβαίνω τον κύριο Αουνίλη που δεν επιλέγεται ένα κβαντικό άλμα. Είναι 200 χρόνια η ιστορία των σιδηροδρομών. Το 1825 ε, κυκλοφόρησε το πρώτο τρένο στην Αγγλία. Κοντεύουν τα 200 χρόνια τώρα επέτειος, χάλιβα με χάλιβα. Μετά από 200 χρόνια, τι τρομακτική αλλαγή θα επιφέρουμε. Η αλλαγή είναι ήρθε ε, με τους ε, τροχούς από καουτσούκ ε, στο μετρό του Παρισιού για πρώτη φορά όταν το είδα αυτό εντυπωσιάστηκα για το πόσο μειώνεται ο θόρυβος και για τους επιβάτες που είναι στην αποβάθρα του μετρό. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν επιλέγετε το κβαντικό άλμα, αλλά γίνεται ένα μικρό βήμα. Δεύτερη ερώτηση. Ε, σε αυτή τη συζήτηση συχνά δεν συζητούμε ένα άλλο είδος θορύβου από το σιδηρόδρομο. Και αυτό είναι όταν ένα τρένο ε, εκτροχιάζεται ε, και ε, και καμιά φορά κάνει και εκατοντάδες μέτρα ε, μέχρι να φρενάρει και να σταματήσει και είναι και αυτό ένα ε, είδος θορύβου που υπάρχει σε εκτροχιασμό τρένων που τρίβεται πια το ο χαλίβας σε άλλα υλικά, σε χαλίκι. Έχω κάνει μια ερώτηση πριν από δυο εβδομάδες για ένα σύστημα ανείχνευσης εκτροχιασμών Υπάρχει ένα σχετικά απλό και φθηνό σύστημα ε, που μπορεί να ενσωματωθεί στα βαγόνια και όταν εκτροχιάζεται ένα τρένο μπορεί πολύ γρήγορα ο μηχανοδηγός ε, να επέμβει και να φρενάρει το τρένο. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην το καταλάβει καν ότι εκτροχιάζεται το τρένο και να συνεχίσει επί χιλιόμετρα ε, να προχωράει ο σειρμός. Ε, πράγμα που και θόρυβο δημιουργεί και καταστρέφει την υποδομή και τα, τα υλικά. Αυτές τι δύο ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Παύλ Τελίτσκα. Uh, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Νίτη, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ήταν σύντομη όπως είπατε, πλην ε, σαφέστατη. Όντως. Μία από τις ερωτήσεις που έχει ήδη απαντηθεί είναι ε, τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος ακριβώς. Θέλω μεγαλύτερες διευκρινήσεις. Εσείς λέτε ότι θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Ε, αυτό ακόμα δεν το έχω καταλάβει πώς θα γίνει και μου λείπει. Μπορείτε λίγο να το διευκρινίσετε. Ευχαριστώ, Πέτερ Λούντγκρεν. Ευχαριστώ. Ε, είχαμε πάει αποστολή στην Φιλανδία και είχαμε συνάντηση εκεί με τους εκπροσώπους των σιδηροδρόμων σχετικά με τα νέα αυτά φρένα από σύνθετα υλικά. Ε, διαπιστώθηκε ότι αποτελούν πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια ε, επειδή παράγεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας και στο χιόνι δεν ε, λειτουργούν καλά. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα ασφαλείας ε, εάν έχουμε νομοθεσία που να καθιστά ε, υποχρεωτικά τα φρένα από σύνθετα υλικά. Ευχαριστώ κύριε Ονιδή για την παρουσίασή σας. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Πρώτη. Προφανώς δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα όσα μας λέτε γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μελετώντας όμως αυτά που μας ζητάτε είναι περισσότερους πόρους και περισσότερα μέσα και εργαλεία, δηλαδή κοινά πρότυπα. Έχω λοιπόν την εξής πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα στο σημείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βλέπω τι μπορούμε να κάνουμε. Παράδειγμα, στην Ευρώπη. ποιε είναι οι πιο κρίσιμε περιοχές για τι οποίε πρόκειται. Δεν μα το έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Έχετε χάρτη για τις οχλήσεις από το θόρυβο συγκεκριμένα. Είναι το πρώτο βήμα για να εργαστούμε από αυτό. Το δεύτερο, ε, ο περιορισμός πρόσβασης ε, για ε, τα βαγόνια που μεταφέρουν εμπορεύματα και κάνουν πολύ θόρυβο από τις ευαίσθητες περιοχές. Ποιες είναι αυτές και πού είναι. Δεν το ξεκαθαρίζετε αρκετά στην έκθεση. Και πώς θα συνδέσετε τώρα τον εξυγχρονισμό ε, των ε, βαγονιών και τη μείωση του θορύβου. Δεν είναι πολύ συμβατά πολλές φορές αυτά. Και ένα θέμα αρμοδιοτήτων επίσης. Ωραία. Περιορισμός του θορύβου. Με προδιαγραφές συγκεκριμένες. Άλλο ισχύει για τη μέρα, άλλο για τη νύχτα. Και πόσες φορές μέσα σε μια χρονιά. Κανονικά η αρμόδια γενική διεύθυνση εδώ είναι η έμβη για το περιβάλλον. Θα συστήσετε κοινή ομάδα εργασία. Σταματώ εδώ, έχω μια σειρά από ερωτήσει ακόμα. Ευχαριστώ η Μαρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση για αυτό το θέμα. Η διαλειτουργικότητα φυσικά είναι σημαντική. Τα προβλήματα μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο συνάδελφος Λούντγκρεν, δηλαδή δεν θα πρέπει τώρα να προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για όλους. Θα πρέπει να αφήσουμε αρκετό περιθώριο στα κράτη-μέλη για εθνικές λύσεις. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία ε, δεν είναι πρόβλημα ο θόρυβος. Τα τρένα κυκλοφορούν μέσα στα δάση. Δεν έχουμε ε, ακούσει ούτε ένα παράπονο, ούτε μία καταγγελία για πρόβλημα θορύβου. Αυτό είναι άγνωστο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όμως αυτό που ζητάτε για τις τεχνικές προσαρμογές. Γιατί ε, όταν φρενάρει το τρένο, αυξάνεται πολύ η απόσταση στην οποία θα σταματήσει. Και δεν ξέρουμε ε, εάν ε, φρενάρει το τρένο με το νέο σύστημα, δεν εκτροχιαστεί. Γιατί έχουμε και πάγο και χιόνι και άλλες συνθήκες ο Πέτερ Λούντκρον γνωρίζει ε, κάλλιστα την κατάσταση και στη Φιλανδία και την Σουηδία. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου μου θύμισε ένας εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι στη Σουηδία χρησιμοποίησαν αυτά τα ειδικά συστήματα ε, πέδησης δοκιμαστικά και πολλές φορές ακριβώς ε, λόγω ε, των καιρικών συνθήκων παραλύει ε, η κυκλοφορία των τρένων το χειμώνα. Ενώ στη Φιλανδία που έχουμε το παλιό σύστημα ε, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Παρόλο που έχουμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, τόσο πολύ χιόνι και τόσο ειδικέ μετεωρολογικέ συνθήκε. Επιμένω λοιπόν να τα λάβει αυτά υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι ίδια η κατάσταση σε όλε τι χώρε, ούτε χωράει ομοιόμορφη και ενιαία λύση. Και όπω ξέρουμε, το καλύτερο συχνά είναι ο εχθρό του καλού. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τι ιδιαίτερε καταστάσει και περιστάσει σε κάθε χώρα και τι συνθήκε που επικρατούν καθώ και τι συνέπειε. Επιπλέον, αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να το είχαμε δει στο τέταρτο ε, σιδηροδρομικό πακέτο. Είναι ένα θέμα ανοιχτό εδώ και πάρα πολύ καιρό και γνωρίζαμε ότι θα το βρούμε μπροστά μας και ότι ήταν προβληματικό. Ισμαήλ Ερτούκ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχής για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία σε τρεις φάσεις ε, δεν είναι αρκετά καλή. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Στην Γερμανία είδε σήμερα ή τουλάχιστον ε, φέτος ε, θα ε, έχουμε μεταξοπλίσει το 50% του τροχαίου υλικού και μέχρι το 2020 θα έχουμε λύσει το θέμα αυτό στην Γερμανία. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλά άλλα κράτη-μέλη δεν έχουν τόσα βαγόνια που πρέπει να μεταξοπλίσουν όσο η Γερμανία και η Γαλλία. αυτή η διαδικασία σε τρεις φάσεις ουσιαστικά προστατεύει ε, κράτη-μέλη που έχουν ε, εκτενείς οδικές μεταφορές και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ε, έχει ασκηθεί πίεση από τα σχετικά λόμπι. Γι' αυτό κύριε Ονίδη θα... Θα ήθελα να μου πείτε πώς προχωράνε τα πράγματα στην ε, Ελβετία σχετικά με την αλλαγή των ραγών. Και επίσης, ε, θα πρέπει να δοθούν ε, κίνητρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε την σχετική διαδικασία και Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται ακόμα στη φάση προβληματισμού ή έχει ήδη ε, διαμορφώσει ένα σχέδιο. Πώς βλέπετε εσείς, ε, πότε πιστεύετε εσείς ότι μπορούμε να περιμένουμε μια συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και επίσης η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, έχει ερωτηθεί σε περίπτωση που επιλέξετε επιδοτήσεις για την ανακαίνιση του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρισκεύσκα. Ε, προφανώς οποιαδήποτε δράση μειώσει το επίπεδο θορύβου και τις ε, συνέπειες του στην ανθρώπινη υγεία θα πρέπει να επικροτηθεί. Ωστόσο, δεν θέλουμε να κάψουμε τα ε, χλωρά μαζί με τα ξερά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, το κόστος, ε, το οποίο νομίζω ότι θα είναι σημαντικό. Αναρωτιέμαι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποιον υπολογισμό σχετικά με την αντικατάσταση των συστηματών πέδησης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Δυτική Ευρώπη σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούνται στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι λοιπόν αρκετά διαφορετικό το επίπεδο κόστους. Δεύτερη παρατήρηση. Νομίζω ότι το κόστος ε, θα ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Έχετε εξετάσει την αναλογία κόστους-όφελους, διότι μπορεί κάποια κράτη να προτιμήσουν να αγοράσουν νέο τροχαίο υλικό αντί να μεταξοπλίσουν το υπάρχον και τι, ε, πώς θα επηρεάσει αυτό την ανταγωνιστικότητα ε, του σιδηροδρομικού τομέα. Αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποια λευκή βίβλος για το θέμα αυτό. Κάποιοι σιδηροδρομικοί οργανισμοί μπορεί να αντιμετωπίσουν τεράστιο κόστος, το οποίο ε, θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητά τους. Ε, αν συγκρίνουμε την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη, και τα διάφορα είδη μεταφορών, σιδηροδρομικές οδικές ε, κλπ. βλέπουμε για παράδειγμα ότι η Πολωνία έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών. Ε, πολλά από αυτά τα χιλιόμετρα όμως βρίσκονται σε αραιά κατοικημένες περιοχές. Ε, δεν υπάρχουν λοιπόν ε, αρνητικές συνέπειες στην ανθρωπινή υγεία λόγω του θορύβου. Να εξετάσουμε λοιπόν τις δυνατότητες όσον αφορά την αντικατάσταση των συστηματών επέδυσης. Θα ήταν χρήσιμο όμως να έχουμε μια λευκή βίβλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα σας τα χαλάσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί ενδείχνεται να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα, να δαπανίσουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να δούμε ε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα μετεξοπλισμού ε, των ε, βαγονιών. Ποτέ δεν έχω λάβει σχετικό email. 12 χρόνια στην Επιτροπή σας συζητάμε τον θόρυβο στο, στους δρόμους, ε, τον θόρυβο στα αεροδρόμια. Κανείς όμως δεν ε, ανέφερε τον θόρυβο ε, στις, στους σιδηροδρόμους. Πρώτα τοποθετήθηκαν οι γραμμές και μετά πήγε ο κόσμος να κατοικήσει κοντά σε αυτές. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα αν κατοικείται δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά νομίζω ότι αυτό αποτελεί ευθύνη των σιδηροδρομικών οργανισμών. Εάν χρειαστεί να γίνει μετεξοπλισμός, Ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ένα πιθανό σύστημα δανείων. Αλλά τα χρήματα αυτά πώς θα διανεμηθούν. Ε? Εγώ είχα διαμέρισμα κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό. Ε, η γραμμή περνούσε στο, ε, δίπλα στον κήπο μου. Ποτέ δεν είχα ακούσει παράπονα. Αλλά βέβαια από ό,τι φαίνεται υπάρχουν παράπονα σε κάποια μέρη. Και συγχωρήστε με, υπήρχε πρόβλημα σε κάποια κρατήδια της Γερμανίας. Εγώ δεν έχω ξανακούσει να υπάρχει σχετικό πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ταπανίσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για τον μετεξοπλισμό ε, συνδρομικών αμαξών. Εάν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, σε περίπτωση που έχουν ιδιωτικοποιηθεί όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, πώς ακριβώς ε, θα γίνει και πόσο μεγάλο μέρος των ε, πόρων αυτών θα είναι επιδοτήσεις. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Εγώ πάντα θεωρώ ότι πρέπει να μετριάζεται ο θόρυβος. Αλλά νομίζω ότι η ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, ανήκει στους σιδηροδρομικούς οργανισμούς. Δεν θα συμφωνήσω με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, που δεν βρίσκω να είναι και τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι τέθηκαν, ε, ότι ακούστηκαν παρατηρήσεις ε, σχετικά με τις διάφορες χώρες. Ε, όπου υπάρχουν ε, εκατοντάδες ε, χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών σε ακατοίκητες περιοχές. Μπορεί παρακαλώ κάποιος να μου δώσει κάποιες απαντήσεις, διότι δεν καταλαβαίνω πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Εγώ πάντως σίγουρα δεν θα στηρίξω μια τέτοια κίνηση. Ευχαριστώ, Ντομινίκ Ρικέ. <coughs> Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο ο Ισμαήλ Αχτούγκ ε, όταν είπε ότι δεν έχουμε μειώσει αρκετά τον κίνδυνο, το θόρυβο συγγνώμη. Διότι όπως ξέρουμε το πρόβλημα είναι ότι λόγω της πολιτικής που ακολουθείται για τους γαλλικούς σιδηροδρόμους έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα δρομολόγια που έχει μειωθεί και ο θόρυβος. Να μια καινοτόμα μέθοδος αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτά τα νέα συστήματα πέδησης που είναι πολύ αποτελεσματικά και έχουν διάφορα ονόματα όχι μόνο είναι κόστος όταν ε, κατασκευάζονται τα βαγόνια αλλά είναι κόστος και κατά τη λειτουργία. Δεν το λέτε αλλά είναι σημαντικό διότι ε, οι ιδιοκτήτες των βαγονιών που συχνά δεν είναι σε δρομικές εταιρείες όταν πρέπει να εγκαταστήσουν αυτά τα νέα συστήματα Μπορούν βέβαια να λάβουν κάποια επιδότηση, κάποια, κάποιο άλλο κίνητρο, αλλά μετά υπάρχουν και έξοδα συντήρησης. Δηλαδή, αυξάνονται και τα λειτουργικά έξοδα. Δεν το αναφέραμε. Τώρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το χρηματοδοτήσει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Και όπως έχει τώρα όμως το κόστος εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων είναι πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, το λειτουργικό κόστο είναι 10% τη επένδυση το χρόνο. Είναι μεγάλο ποσοστό. Τι θα γίνει λοιπόν. Είναι πολλά τα ποσά, τα, τα που θα πρέπει να δαπανίσουμε για να συντηρούμε τα βαγόνια που θα επανεξοπλιστούν με τους νέους μηχανισμούς αυτούς. Πρόεδρος. Ναι, τώρα να σχολιάσω κι εγώ. Δεν θα σας εκπλήσει βέβαια. Αυτή τη συζήτηση την ξεκινήσαμε πριν από 10-12 χρόνια. Α, με συγχωρείτε, δεν σα είδα. Ναι, βέβαια, θα σας δώσω μετά το λόγο. Θυμάμαι ότι τότε ήμουν ο μόνος. Αλλά έκτοτε έχουν αλλάξει τα πράγματα και υπάρχει πλειοψηφία και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο για αυτή την προσπάθεια. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Επιτύχαμε να υπάρχει χρηματοδότηση για το τροχαίο υλικό, ήταν δύσκολο το επιβάλαμε. Και τα βρήκαμε και 1%, 260 εκατομμύρια από τον προπολογισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό μπορούν ε, να κάνουν αίτηση γι' αυτό τα κράτη ή οι επιχειρήσεις. Πού υπάρχει σύγκρουση. Αλλά κανείς δεν ανησυχεί για τα 10 δισεκατομμύρια που επενδύονται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να φτιάξουμε αυτά τα τείχη κατά μήκο των γραμμών. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να μένω γύρω ε, πίσω από έναν τείχο. Θέλω να βλέπω γύρω μου. Δέκα δις έχουμε δώσει για αυτούς τους Τι θα θέλαμε για να επανεξοπλίσουμε τα νέα βαγόνια είναι επίση σαφέ. Ούτω ή άλλω θα πρέπει να έχουν αυτού του νέου μηχανισμού. Τεχνικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μόνο πολιτική βούληση για να το εφαρμόσουμε. Και για την ε, μεταφορά εμπορευμάτων που κατά πάνω από 50% είναι διαμεθοριακή μεταφορά, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή λύση. Γιατί οι εθνικέ λύσει δεν επιβάλλουν τίποτα, εφόσον είναι διασυνοριακέ αυτέ οι μεταφορέ. Τι θα κόστιζε λοιπόν για να αλλάξουμε 80% των βαγονιών, πόσο θα μα κόστιζε, 1,2 δι. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει 8,8 δις γιατί δεν θα αντιμετωπίζαμε μέσω τείχων το θόρυβο, αλλά θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα στην ε, πηγή. Η Ελβετία θα το έχει μέχρι το 2020 και πάρα πολλά περνάνε από την Ελβετία. Μπορούμε να πούμε σε επιχειρήσεις, ε, κοιτάξτε να δείτε, δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα αυτά, αλλά δεν θα μπορείτε να περάσετε από την Ελβετία. Και επειδή πολλέ φορέ το κόστο ακόμη για τα αυτοκίνητα είναι υψηλό στην ε, Ελβετία, περνάνε όλοι από την Αυστρία. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα το ανεχθούν για πολύ καιρό η Αυστρία. Έχουμε λοιπόν τι δυνατότητε, θα κάνουμε εξοικονομήσει και χρόνο και θα έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Είναι μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν. Αλλά μια τέτοια κατάσταση είναι φαίνεται στην πολιτική είναι το δυσκολότερο να την επιβάλλει. Αλλά σα παρακαλώ να υποστηρίξουμε την Κομισιόν. Στη Γερμανία το έχουμε πει κατά 50%. Θυμάμαι πριν από 5-6 χρόνια όταν είχαμε αυτή τη συζήτηση, μα λέγανε ότι μόνο μια επιχείρηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να τα επιβάλλουμε τόσο γρήγορα. Αλλά ακόμη και οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι δεν συμφωνούσαν. Εν μεταξύ υπάρχουν πολλέ επιχειρήσει και δημιουργήθηκαν και πολλέ θέσει εργασία. Και ανθίζει ο κλάδο. Ανθεί ο κλάδο. Και κανεί πριν από πέντε χρόνια δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε επιτύχει σε πέντε χρόνια και το επιτύχαμε. Δείξαμε λοιπόν ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Και φυσικά ο σημαντικότερος διάδρομος ε, για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι Ρότερνταμ Γενέβη και ε, Γένοβα συγγνώμη και ε, αυτό το, κάθε τρία λεπτά περνάει ένα τρένο από αυτόν τον διάδρομο και ο θόρυβος σε ορισμένα σημεία είναι πραγματικά απίστευτος και αφόρητος και πολλοί όταν το διαπίστωσαν ε, κατάλαβαν τι είναι το πρόβλημα και σε ορισμένε περιοχέ δεν μπορεί κανεί να κοιμηθεί. Ορισμένοι νόμιζαν ότι ορισμένε περιοχέ ε, θα εξακολουθούσαν να είναι τουριστικέ, αλλά πλέον έχει καταστραφεί ο τουρισμό του. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσει. Μερικού ε, μπορεί να του πειράζει ο θόρυβο, ακόμη και αν κοιμάσαι δίπλα σε ένα τρένο. Εγώ όμω δεν είμαι από αυτού. Και είπα ότι οι, οι συνδρομικέ μεταφορέ έχουν μέλλον μόνο εάν το λύσουμε σύντομα το πρόβλημα αυτό εντάξει, και εγώ ίδιος για την πολιτική μεταφορών συχνά επικρίνω τη Γερμανία. Αλλά σε αυτό το σημείο, στην ε, κυβερνητική συμφωνία στη Γερμανία, λέγεται ότι μέχρι το 2020 πρέπει να γίνει. Και εγώ καταλαβαίνω ότι και η συντήρηση έχει ένα κόστος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ε, δεν θα χρειάζεται να ε, φρενάρετε απότομα, θα φρενάρετε πολύ πιο σταδιακά και αυτό θα μειώσει το κόστο συντήρησης. Μπορεί τώρα να είναι κάπως πιο ακριβά γιατί πρέπει να γίνει επένδυση για να υπάρξει αυτή η μετατροπή αλλά ε, μακροπρόθεσμα όλοι κερδίζουν και οι επιχειρήσεις ε, και ο τουρισμός ε, και η ύπεθρος και όλοι όσοι ζουν κοντά για όποιος κοιμάται καλά μπορεί να εργαστεί καλά είναι πιο παραγωγικό. Συνολικά λοιπόν είναι μια επένδυση που θα ωφελήσει και τους πολίτες αλλά και τον κλάδο και φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος και τις συνδρομικές μεταφορές, γιατί θα γίνει ε, ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον ε, ε, η μεταφορά εμπορευμάτων. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να είναι πιο φιλόδοξη, να θέσει ως στόχο το 2020 και να έχουμε στις ε, χώρες διαφοροποιημένη πολιτική κόστους χρήσης των συνδρομικών γραμμών. Όποιος κάνει περισσότερο θόρυβο, με βάση την αρχή ο Μολύνο πληρώνει, πρέπει να πληρώνει περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να το εφαρμόσουμε συγκεκριμένα αυτό. Και τώρα ε, και η κυρία Βίλκουν και μετά ο κύριος Λούντγκρεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε προσοχή στο θόρυβο Ε, τρένων, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα των σιδηροδρομικών οργανισμών, των διαχειριστών του δικτύου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάνει και τον ε, χωροταξικό και πολυδομικό σχεδιασμό και που θα χτίσουν. Και όταν περιορίζεται ο θόρυβος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ε, που να συμφέρει οικονομικά. Ξέρουμε ότι δεν είναι παντού μεγάλο πρόβλημα ο θόρυβος σε όλες τις περιοχές. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε εθνικά προγράμματα ε, αντικατάστασης ε, των μηχανισμών πέδησης των βαγονιών. Ελπίζω να καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στις βορειοευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους συστήματα πέδησης. Στις σκανδιναβικέ χώρες τα έχουμε δοκιμάσει. Ξέρετε, ο χειμώνα είναι πάρα πολύ ε, βαρύς και σφοδρός, με χιόνι και πάγο ε, που ε, παγώνουν αυτά τα συστήματα πέδησης τα οποία δεν μπορούν να φρενάρουν μετά ή χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη απόσταση για να φρενάρουν, μειώνεται η ασφάλεια. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και θέλω να βεβαιωθώ ότι το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πήγε αντιπροσωπεία μας στη Φιλανδία το Φεβρουάριο και με τρένο ταξιδεύαμε και μας τα είπαν οι εμπειρογνώμονες ότι είναι πρόβλημα αυτό για τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Και ανησυχούν πάρα πολύ για τα σχέδια αυτά γιατί γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στις βορειοευρωπαϊκές και σκανδιναβικές χώρες. Και είναι θέμα ασφάλειας πλέον. Ευχαριστώ και πάλι ο Πέτερ Ευχαριστώ. Ναι, συμφωνώ φυσικά με τους συναδέλφους από τη Φιλανδία. Ε, τα φρένα από σύνθετα υλικά είναι πολύ καλά όταν λειτουργούν, αλλά δεν λειτουργούν παντού και δεν ε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο βορρά εφόσον δημιουργούν πρόβλημα ε, ασφαλείας. Και στη Φιλανδία και στη Σουηδία έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέπετε τουλάχιστον ε, κάποια παρέκκληση για λόγους ασφαλείας. Πρόεδρο, σε μία σύντομη παρατήρηση, προτού να σας δώσω το λόγο 30 δισεκατομμύρια δώρο παίρνουν ε, οι αερομεταφορείς ε, από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο διότι δεν πληρώνουν φόρο επί της κυροσύνης. Ε, αλλά εάν δεν έχουμε ευρωπαϊκή λύση, επιλέξουμε εθνικές λύσεις και η Γερμανία πει ότι μέχρι το 2020 τέλος, τότε το 80% των εμπορευματικών αμαξών θα πρέπει ή να μεταξοπλιστεί ή δεν θα επιτρέπεται πια να ε, ε, ε, να λειτουργούν. Οπότε δεν αποτελεί επιλογή να κλείσουμε τα μάτια και να μην κάνουμε τίποτα. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους Ευρωβουλευτές για τις παρατηρήσεις τους. Οι απόψεις που ακούστηκαν αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Νομίζω ότι οπωσδήποτε πρέπει να επιλέξουμε ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα αυτό, διότι αλλιώς ε, δυστυχώς θα καταλήξουμε σε πολύ περίπλοκες καταστάσεις, όπως ε, βλέπουμε στις περιπτώσεις των αεροδρομίων και των οδικών μεταφορών. Μέχρι τώρα καταφέραμε να διατηρήσουμε την ε, ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς παρά διάφορες προσπάθειες ε, κρατών μελών ε, και ε, τοπικών αρχών να επιβάλλουν απαγορεύσεις. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε εσωτερική αγορά στον ε, σιδηροδρομικό τομέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προωθήσουμε τις εμπορευματικέ μεταφορές ε, στους σιδηροδρόμους. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για να ε, αποφύγουμε να εμφανιστούν νέα εμπόδια που θα μειώσουν τις δυνατότητες για τον τομέα αυτόν. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και γι' αυτό ακριβώς εξετάζουμε τον πιο οικονομικό τρόπο να ε, επιλύσουμε το πρόβλημα και αυτό είναι ο λόγος που η αξιολόγηση αντικτύπου εξετάζει το κόστος ε, μεταξοπλισμού ε, σε σύγκριση με άλλες λύσεις όπως είναι το κόστος συντήρησης και η κατανομή του κόστους σε όλο τον κύκλο ζωής του στόλου καταλήξαμε ότι είναι καλύτερο να έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον μεταξοπλισμό ε, του συνόλου των ε, αμαξών, διότι χρησιμοποιούνται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ δύσκολο να περιορίσουμε την χρήση κάποιων αμαξών σε συγκεκριμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόβλημα θορύβου. Τούτου λεχθέντος, ε, όλες οι παρεμβάσεις σας ε, αποτελούν αιτήσει για αναλογικότητα. Εάν ε, τα νέα φρένα από σύνθετα υλικά αποτελούν πρόβλημα ασφαλείας, θα προβλέψουμε παρεκκλήσεις. Έχω ακούσει το πρόβλημα, όπως και εσείς άλλωστε. Δεν έχω λάβει όμως τα αποδεικτικά στοιχεία, ούτε Έχω δει ε, κάποια άλλη παρουσίαση που να μου δείχνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ακραίες καιρικέ συνθήκες. Αν όμως ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο θα το λάβουμε υπόψη μας και θα φροντίσουμε η υποχρέωση με το εξοπλισμό να συνοδεύεται και από κάποια δυνατότητα παρέκκλησης. Νομίζω μια άλλη παρέκκληση που θα πρέπει να είναι δυνατή αφορά το χρονοδιάγραμμα. Και θα βασίζεται στο αν ε, επηρεάζονται πολίτες από το θόρυβο ή όχι και το αν μπορεί να περιοριστεί η χρήση συγκεκριμένων αμαξών σε ε, συγκεκριμένες περιοχές. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω συνομιλίες μαζί σας ε, και με τις εθνικές αρχές. Θα εξετάσουμε το πρόβλημα. Έχουμε χαρτογραφήσει τις ε, ευαίσθητες περιοχές ε, και θα παρουσιαστούν οι σχετικοί χάρτες ε, στο Ρότερνταμ στο πλαίσιο του TNT των Ευρωπαϊκών Δικτύων. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα συστήματα πέδησης από σύνθετα υλικά. Ναι, υπάρχουν εναλλακτικές. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε ε, ε, στους ε, τείχους για την μείωση του θορύβου, που βέβαια είναι δαπανηρή. Δεν έχουμε σταματήσει την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Τα εξετάζουμε όλα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος Shift to Rail μεταφορά στους σιδηροδρόμους δηλαδή. Και εξετάζουμε τι μπορεί να μειώσει τον θόρυβο στα βαγόνια αλλά και στις υποδομές. Στις υποδομές ε, υπάρχει η δυνατότητα του grinding, κάτι που επιτρέπει καλύτερη απορρόφηση του θορύβου που παράγεται με ε, συγκεκριμένα μέτρα στις σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά δυστυχώς δεν αρκεί. Γι' αυτό θεωρούμε ότι τα νέα συστήματα απέδησης ε, αποτελούν ε, απαραίτητη λύση. Επίσης, τέθηκε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Θα χαρώ πολύ μετά από τη σημερινή συζήτηση και τις συζητήσεις που έχουμε με τις εθνικές αρχές να σας υποβάλω κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τα μέσα που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε. Όσον αφορά το συνολικό χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το 2020 ε, που συμπεριλαμβάνεται στην ε, απόφαση της Ελβετίας. Ε, ανάλογη ημερομηνία αναμένεται από πλευράς της Γερμανίας. Ελπίζουμε λοιπόν σύντομα να έχουμε μια ημερομηνία για την ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να ευθογραμμιστούν όλοι και να μην έχουμε πρόσθετα προβλήματα. Θα συμπεριλαμβάνονται βέβαια δυνατότητες παρέκκλησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Για παράδειγμα, το κατά πόσο επηρεάζεται ο πληθυσμός ε, ή όταν υπάρχουν ε, ε, κίνδυνοι ή προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια. Κύριε Βαντενκάμπ, μία πολύ σύντομη περίληψη των μέτρων έχετε που αντικατοπτρίζει τα μέτρα της Κομισιόν, ε, το αποτέλεσμα της μελέτης αντικτύπου και τις προθέσεις ε, που ε, εξέφρασε ο Επίτροπος προσωπικά. Κατά την διάσκεψη για το TNT, τα διευρωπαϊκά δίκτυα στο Ρότερνταμ, θα έχουμε και μια διακήρυξη ε, που θα αντικατοπτρίζει τη συνένεση του τομέα, όχι μόνο όλων των χωρών, αλλά και όλων των άλλων παραγόντων, όλων των άλλων φορέων ώστε να προχωρήσουμε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μεταξοπλισμό όλων των τρένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Um, λοιπόν, μια στιγμή. Κάτι ξέχασα ε, να απαντήσω, ναι, είναι σημαντικό. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ήδη από τώρα είναι να κοιτάξουμε μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για ευρύτερη χρηματοδότηση σε ε, αυτή την περίπτωση για το θόρυβο. Σε σχέση λοιπόν όμως με όλα αυτά, όντως έχουμε αρχίσει τη συζήτηση με τους ε, συναδέλφους από διάφορες υπηρεσίες, όχι μόνο Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, έτσι ώστε είτε να ε, ε, βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε απόσυρση, είτε να δούμε πώς μπορούμε να εθαρρύνουμε ε, κάτι σε ευρωπαϊκό και όχι πλέον εθνικό επίπεδο. Αυτό δεν αφορά μόνο το θόρυβο, αλλά θα ήταν πάρα πολύ θετικό και για την ασφάλεια γενικότερα, αλλά και για το περιβάλλον, διότι θα επέτρεπε ακριβώς ε, όλο αυτό το υλικό να ανακυκλώνεται με τρόπο ολοκληρωμένο και με σεβασμό στο περιβάλλον. Να βοηθήσει και τη βιομηχανία μας να έρθει πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες και πολύ πιο γρήγορα. Η ιδέα υπάρχει, δεν μπορώ να σας δώσω χρονικό ορίζοντα, ούτε ε, επίσημα και στοιχεία. Είναι πολύ περίπλοκο και είναι και πάρα πολύ πρώιμο το στάδιο, να σας πω. Ο Πρόεδρος. Λοιπόν, τώρα δυστυχώ θα πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, για τις απαντήσεις, ερωτήσεις και βεβαίως το θέμα θα συνεχίσει να μας απασχολεί και ερχόμαστε στο επόμενο σημείο για την ομάδα δράση για τον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αρχίσει η επόμενη συζήτηση και αν δεν σας ενδιαφέρει παρακαλώ να αποχωρήσετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα σε μέρη σε διάταξη που αριθμό 13. Σωρίζω θερμά την ομάδα δράση για τον τουρισμό στη σημερινή μας συνεδρίαση. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το Μανιφέστο για τον τουρισμό, πρόγραμμα δράσης, ε, που έχουν εκπονήσει από κοινού ιδιώτες και δημόσιοι φορείς. Έχει διανεμηθεί το μανιφέστο και υπάρχουν και αντίγραφα εδώ στην αίθουσα. Πριν παρακαλέσουμε τους εμπειρογνώμονες να μας το συστήσουν, θα τονίσα ότι ε, καλωσορίζω πραγματικά αυτή την πρωτοβουλία. Η συνθήκη της Λισαβόνα ε, ορίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στην Ευρώπη, άρα χρειάζεται συντονισμένη δράση οπωσδήποτε των φορέων και αξίζει υποστήριξη. Επίσης, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι τα πεδία δράση του μανιφέστου σε μεγάλο βαθμό καλύπτουν τις προτεραιότητες που παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2015 η Επίτροπο στη Μαδρίτη και γι' αυτό αναμένονται συνέργειες για την υλοποίηση ε, του μανιφέστου. Μερικές από τις ε, ενέργειες αυτές και τα, τις δράσεις και τα μέτρα συζητήσαμε και στο παρελθόν, ας πούμε πώς θα ξεπεραστεί η ε, εποχικότητα του τουρισμού και πώς θα είναι πιο προσβάσιμη η τουριστικοί ε, προορισμοί. Τον Οκτώβριο εγκρίναμε και έκθεση πρωτοβουλία τη συναδέλφου Ζαπέλα Ντεμόντε, που ασχολήθηκε με τι ιδιαίτερε προκλήσει ε, του κλάδου του τουρισμού, που βλέπουμε και στο μανιφέστο, όπω είναι η ψηφιοποίηση ή ε, ο αηφόρο και βιώσιμο τουρισμό. Τώρα όμως θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρο της ομάδα, τον κύριο Ισφαν Ουχέλη, ο οποίος εκπώνησε και αυτός ε, την έκθεση μαζί με άλλους συναδέλφους και δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης για τη δυνατότητα που μου δίνετε για να σας παρουσιάσω αυτή την ε, διακήρυξη αρχών με την παρουσία των ε, φορέων που συμμετείχαν στην εκπόνησή του, στην εκπόνησή της και Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία της Επιτροπής μας για τη, βοήθεια, για που μου έδωσαν κατά την προσπάθεια αυτή. Η προσπάθεια η οποία έχει στόχο να δημιουργήσουμε μια εντελώς νέα κατάσταση προς το συμφέρον όλων όσων ασχολούνται με τον τουρισμό. Και ελπίζω να μας υποστηρίξετε και στην προσπάθεια που κάνουμε για να υπάρξει διοργανικός διάλογος και διάφορες περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να ε, λάβουν χώρα εδώ στο Κοινοβούλιο και μέσω του Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη βοήθειά σας, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θέλω να τονίσω ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ στην αίθουσα Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κλάδο αυτόν γιατί είναι ένας κλάδος ε, που απασχολεί πολλά εκατομμύρια εργαζόμενους. Είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους ε, της οικονομίας μας και γι' αυτό πιστεύω ότι στο μέλλον τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να ε, προωθήσουν περισσότερο από ό,τι μέχρι στιγμής τα συμφέροντα του κλάδου αυτού. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για το ότι διάφοροι φορείς του κλάδου αυτού για πρώτη φορά προσπαθούν να δημιουργήσουν, να εκπονήσουν ένα κοινό πρόγραμμα δράσης και μια κοινή διακήρυξη αρχών. Αυτό πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα θετικό και το χαιρετίζουμε και πρέπει να το στηρίξουμε. Είναι πολύ σημαντικό και χαιρόμεθα που σημαντικοί φορείς και σημαντικοί ε, εμπειρογνώμονες και ειδικοί μπορούν να συζητήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα και θα έπρεπε να έχουμε τακτικά τέτοια δυνατότητα. Θέλω καταρχάς ε, να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Αρκεί απλώς ένα μανιφέστο, μια διακήρυξη αρχών. Αρκεί να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το στο Κοινοβούλιο. Όχι, σίγουρα δεν επαρκούν όλα αυτά. Γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα. Μόνο και μόνο μια διακήρυξη και μια τέτοια συζήτηση. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, όλοι οι βουλευτές ευρωβουλευτές δηλαδή, και διάφοροι άλλοι που ε, ενεργά θέλουν να εφαρμοστεί αυτή η διακήρυξη ε, αρχών, πρέπει να συνεργαστούμε, να συνδυάσουμε τις ενέργειές μας. Διότι συχνά ακούμε ότι υπάρχει πολλή ανεργία στην Ευρώπη. Και τονίζουμε ότι θέλουμε να υπάρξει επαναβιομηχάνηση της ε, Ευρώπης. Δεν μπορούμε λοιπόν, εφόσον τα λέμε όλα αυτά, να διαπιστώνουμε ότι στο πρόγραμμα Juncker και σε άλλα προγράμματα δράσης ούτε καν αναφέρεται ο τουρισμός. Ενώ ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους, όπως είπα, από πλευράς απασχόλησης. Και έχει πολλές δυνατότητες δημιουργίας περαιτέρω θέσεων απασχόλησης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε τόσα εκατομμύρια νέους εργαζόμενους από την Ισπανία μέχρι την Ουγγαρία. Πολλοί νέοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Και τα συστήματα εκπαίδευσής μας δεν ασχολούνται επαρκώς με τις δυνατότητες κατάρτισης νέων ε, για τον τουρισμό, όπου είναι πολύ απλό για νέους να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Ακούμε επίσης και διαπιστώνουμε ότι ε, ο τουρισμός είναι βεβαίως μια υπηρεσία και άρα δεν είναι βασικός ε, κλάδος οικονομικής δραστηριότητας. Υποτιμάται έτσι. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, πιστεύω, ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο ε, υπηρεσία. Νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ πιο βασικός κλάδος της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και περισσότερες συγκεκριμένες συνεργασίες και εταιρικέ σχέσεις στον κλάδο αυτό. Τα κράτη-μέλη επίσης δεν θα πρέπει να θυσιάζουν τον τουρισμό για διάφορες ε, σκοπιμότητες ή για διάφορες ε, συγκρούσεις για θέματα αρμοδιοτήτων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η υποστήριξη του τουρισμού είναι κάτι το αναγκαίο για όλους μας, για όλα τα κράτη-μέλη, όπως βέβαια και για άλλους τουριστικούς προορισμούς. Και αν το κάνουμε αυτό, πραγματικά θα έχουμε πολύ σύντομα σημαντικά αποτελέσματα. Με αυτά τα εισαγωγικά θα ήθελα τώρα να δώσουμε το λόγο σε εκπροσώπους 7 ειδικών οργανώσεων. Δεν ήταν απλό να επιλέξουμε αυτούς τους 7. Είχαμε 13 οργανώσεις, 13 φορείς το πιο σημαντικό όμως είναι να μπορέσουμε να ακούσουμε ε, ε, καινοτόμες προτάσεις για αυτά. Ευχαριστώ Ιστβάν. Έχουμε λοιπόν ε, προσκαλέσει έξι εμπειρογνώμονες. Ο χρόνος είναι περιορισμένος φυσικά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο των έξι λεπτών. Ο πρώτος είναι ο Εδουάρδο Σανταντέρ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων, ETC, European Travel Commission. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτές. Ε, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω μία μοναδική πρωτοβουλία στην ιστορία του τομέα τουρισμού στην Ευρώπη. Ο τουρισμός ε, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, ε, αντιπροσωπεύει το 5% του ΑΕΠ και συμβάλλει συνεισφέρει 25 δισεκατομμύρια ευρώ στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, προωθεί την πολιτιστική κληρονομιά, την, ε, τις υποδομές ε, και επίσης την ευρωπαϊκή συνείδηση. Η Ευρώπη παραμένει ο υπαριθμός ένα τουριστικός προορισμός σε όλο τον κόσμο, ωστόσο χάνει σε ανταγωνιστικότητα. Ε, άλλες περιοχές του κόσμου, δημιουργούν ε, περιβάλλον πιο κατάλληλο να ε, υποδεχτεί όλο και περισσότερους ταξιδιώτες. Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον συνολικό αντίκτυπο του τομέα και τον μεγάλο αριθμό των ενδιαφερόμενων κύκλων. Συμπεριλαμβάνονται οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι εταιρείε ε, αερομεταφορών ε, και χερσαίων μεταφορών, ε, τον τομέα εστίασης, τον τομέα ψυχαγωγίας και πολλούς άλλους. Σήμερα Θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι έχουν συνεργαστεί ε, για να εκπονήσουν ε, το μανιφέστο που τονίζει τις προτεραιότητες ε, για τον ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα τα επόμενα χρόνια. Πάνω από 30 ενώσεις συμμετέχουν και συμμετέχουν και ιδιωτικοί και δημόσιοι φορεί. Ε, καλή διακυβέρνηση, ψηφιοποίηση του τομέα, πρόθεση της Ευρώπης ως τουριστικό προορισμό, ε, βελτίωση των ε, δεξιοτήτων και καλύτερε διασυνδέσει αποτελούν προκλήσεις του τουριστικού τομέα σήμερα. Και θέλουμε αυτές τις προκλήσεις να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες είναι ώρα να συνεργαστούν οι διάφοροι φορείς του τομέα ε, και να ακουστεί η φωνή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε λοιπόν πολύ σήμερα που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ε, το μανιφέστο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όπως ε, αναφέρθηκε ε, από την Επίτροπο Βιανκόφσκα στην ε, δήλωσή της εδώ σε τούτη την Επιτροπή, θα πρέπει να εντοπίσουμε προτεραιότητες εφικτές για τον τομέα μέσα στους επόμενους μήνες. Σήμερα θα σα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες αυτές τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τη οποία είμαι πρόεδρος ο τουρισμός ε, αποτελεί ε, σημαντικό εργοδότη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πρωτού να κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία της Επιτροπής Τραν, της Επιτροπής, τη γραμματεία της ομάδας της πρωτοβουλίας μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Χέιλι που επέστε την προσοχή της Επιτροπής σας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενο ο Τιμ Φέχεστ από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ροπερέτο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, όπω ακούσαμε, η συνθήκη τη Λισαβόνα, όπω το λέει και το 2010 η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μα επιτρέπεται εξή πρόθεση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος, ενθάρρυνση της συνεργασίας κρατών μελών, κυρίως με την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών ε, και βελτίωση της προσέγγισης στο τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη και ε, τον τουρισμό στις υπόλοιπες πολιτικές. Δηλαδή ζητούμε ένα νέο πρόγραμμα δράσης που να βασίζεται σε αυτούς τους τομείς όπου έχει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρμοδιότητες, ενιαία αγορά, διαβατηρίων, ε, περιβαλλοντικές διατάξεις. Χρειάζεται μια εγκάρσια, όπως ακούσαμε, προσέγγιση, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως ε, η κατάσταση και να δημιουργηθεί η οικονομία που ζητεί η συνθήκη με τις θέσεις εργασίας που μας χρειάζονται. Ε, δεν θα ε, χρειαστεί υπερβολική φυσικά ρύθμιση ούτε ε, επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τουρισμό στη δημιουργία θέσεων εργασία. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή τουρισμού και όπου οι αρμοδιότητες παραμένουν εθνικές ή περιφερειακές, θα μπορούσε να χαρτογραφήσει ε, την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιμείνει ε, στην ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Εδώ ε, έχουμε θέματα ιδιοκτησίας, ανέγερση κατοικιών, φορολογίας κλπ. Υπάρχουν και διάφορες μορφές εργασίας στο τουρισμό, όπως είναι εποχιακή εργασία, αυτοαπασχολούμενοι, πολλές φορές είναι πολλά τα εμπόδια. Ε, ε, χάνονται και ε, φορολογικά έσοδα για το κράτος, εποφελείται η παραοικονομία και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες θα πρέπει να ενισχυθούν και δεν θα πρέπει να τιμωρούνται ή να αποθαρρύνονται όταν καινοτομούν ή έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα και σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις θέλω να αναφέρω κάτι που δεν λέει το μανιφέστο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα έτσι ώστε να έχουμε συντονισμό και δημοσίευση πληροφοριών από ε, τις αρμόδιες ε, κρατικές αρχές για απειλές τρομοκρατικές, προβλήματα δημόσιας υγείας και άλλα γενικότερα θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό. Θα πρέπει να έχουμε ταχεία ενημέρωση σε πολλές γλώσσες η αγορά παγκοσμίω διψάει για ε, την πληροφορία που δεν έχουν οι ε, αρμόδιοι ε, του κλάδου και βεβαίως οι διάφορες υπηρεσίες έχουν άλλη δουλειά από το να ενημερώνουν για το τι γίνεται σε διάφορες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερική η Ιαπωνία κτλ. Χρειάζεται οπωσδήποτε ταχεία ενημέρωση ε, για να υπάρχει μια εύρεθμη λειτουργία της αγοράς και να μην έχουμε ε, υπερβολικές αντιδράσεις. Ε, τι είναι ο τουρισμός, πώς θα αναπτυχθεί, είναι οι θέσεις εργασίας που μας ενδιαφέρουν, το παγκόσμιο μερίδιο ε, πώς το μετράμε, τη δαπάνη, τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, ε, τι παράγει ο τουρισμός, τι εξάγει, τι εισάγει. Είναι η γνώμη των καταναλωτών. Θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να τους ρωτήσουμε και εκείνους, να ρωτήσουμε και τις διάφορες τοπικές κοινότητες. Με δύο λόγια θα πρέπει να αναπτύξουμε δείκτες επιδόσεων που να ταιριάζουν με τους στρατηγικούς στόχους και χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση, περισσότερα στοιχεία και καλύτερα και ποιοτικά και ποσοτικά. Τίθενται και τα θέματα της χρηματοδότησης. Ε, θα πρέπει τα έργα μας να ακολουθούν τα λόγια μας. Και αν πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον τουρισμό, ιδιαίτερα για του νέου, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουν και επενδύσει η χρηματοδότηση που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φτάσει στους στόχους της συνθήκης είναι ελάχιστη. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, μεγάλα ποσά για τις μεταφορές και θα επηρεάσουν θετικά το τουρισμό, θα αναπερθούν οι συνάδελφοι. 11 είναι οι πηγές ε, ε, χρηματοδότησης, αλλά καμία δεν είναι ειδικά για τον τουρισμό. Ούτε έχει εντολή υπάρχει μια περιοδική δημοσίευση ε, των ποσών που ε, διατίθεται για τον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να αξιολογείται σωστά. Θα πρέπει λοιπόν πέρα από ε, τα κανονιστικά, τα φορολογικά θέματα ή τις των διαβατηρίων, να κάνουμε μια προσπάθεια με τη σωστή χρηματοδότηση για να πιάσει τόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χριστιαν Hospitality Europe. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί κύριοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, όπως όλοι ξέρουμε, ο τουρισμός γίνεται όλο και σημαντικότερος για την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί είναι ένας από τους λίγους τομείς που εξακολουθεί να δημιουργεί θέσεις εργασίας και συμβάλλει ουσιοδό στην ανάπτυξη. Παρά τα ανεπανάληπτα χαρακτηριστικά της Ευρώπης, που έκανε την αύξηση του τουρισμού πολύ σημαντική στην Ευρώπη εξακολουθεί να χάνει τμήματα της αγοράς παγκοσμίω. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που μειώνουν την ανταγωνιστικότητά του. Πρώτον πρέπει να αναθεωρήσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για να μειωθεί η γραφειοκρατία και το φορολογικό βάρος. Το φορολογικό και διοικητικό πλαίσιο για τον τουρισμό έχει να κάνει με ασυντόνιστη εφαρμογή των φόρων και δασμών σε ευρωπαϊκό, τοπικό και κρατικό επίπεδο δημιουργεί ασυνέπειες και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Για να αποτιμήσουμε τον αντίκτυπο της φορολόγησης στον τουρισμό, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως λέει και η έκθεση Ντεμόντε, να υπάρξει μια έκθεση που να καταλήξει σε συγκεκριμένα πορίσματα για να υπάρξει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Δεύτερον, Πρέπει να αξιολογήσουμε την οικονομική και κοινωνική επίπτωση από την ε, οικονομία διανομής. τη συμμετοχική οικονομία. Να δούμε τι θετικά έχει αυτό για την ε, προστασία των καταναλωτών. Η επέκταση της συμμετοχικής οικονομίας μπορεί να βοηθήσει και τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας μειώνοντας ε, την αδήλωτη και παρά, παράτυπη εργασία. Όπως ζητάει και η εκθεσή Ντεμόντε, μια τέτοια μελέτη θα μας ε, δώσει και τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Τρίτον, να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές από την Ένωση για να εφαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία για τη συμμετοχική οικονομία για να υπάρξουν θεμητές συνθήκες ανταγωνισμού για όλα τα θέματα. Το μανιφέστο χαιρετίζει την έκθεση Ντεμόντα για άλλη μια φορά που τονίζει ότι για να υπάρξει προστασία των καταναλωτών οι κανονισμοί για την υγεία και ασφάλεια που ισχύουν για την παραδοσιακή τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να ισχύουν και για τη συμμετοχική οικονομία. Τέταρτον, να υπάρξει διαφάνεια και ουδετερότητα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσω του ίντερνετ. Τα αποτελέσματα ερευνών, search στο ίντερνετ, θα πρέπει να είναι στην αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για του καταναλωτέ. Ο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έρευνε στο ίντερνετ για να βρει αποτελέσματα είναι πολύ βασικέ για τι αποφάσει που παίρνουν οι καταναλωτέ. Οι μηχανέ ε, αναζήτηση θα πρέπει να είναι ουδέτερε. Όλα τα θέματα που αφορούν την διαφήμιση πρέπει να αναφέρονται σαφώς και να εξηγούνται, όπως ε, κατέδειξαν διάφορες μελέτες. Πολλοί καταναλωτές κάνουν κλικ επί των αποτελεσμάτων που θεωρούν ότι τους είναι πιο χρήσιμα. Ο τρόπος παρουσίας των αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να παραπλανεί τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ πολύ ε, στην προσπάθεια να επιλύσουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή είναι ο Άνταμ Ποτόρα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ε, κύριοι Ευρωβουλευτέ. Η Επιτροπή σας είναι η Επιτροπή Μεταφορών, οπότε μάλλον ε, μιλάτε κυρίως ε, για προβλήματα και προκλήσεις του τομέα μεταφορών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα δίκτυα μεταφορών στην Ευρώπη είναι πολύ καλά ε, αναπτυγμένα σε σχέση με το υπόλοιπο του κόσμου και ε, μπορούν ε, να αποτελέσουν μοναδικό ατού στον, στην αγορά τουρισμού. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δεν εκμεταλλευόμαστε όλες τις δυνατότητες. Δυστυχώς, όταν μιλάμε για ταξίδια μακρινά, ε, συχνά ε, τα πάμε χειρότερα από τις ΗΠΑ που είναι απόλυτα επικεντρωμένες ε, στα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, εάν θέλω να πάω από τη Νέα Υόρκη στο Σικάγο, μπορώ να κλείσω ένα εισιτήριο τρένου. Εάν θέλω να πάω από τις Βρυξέλλες ε, στην ε, δική μου πόλη, την Βουδαπέστη, 1400 χιλιόμετρα, ε, δεν μπορώ να κλείσω με μια το εισιτήριο για όλη τη διαδρομή. Και αν έχω την τρελή ιδέα να πάρω μαζί μου το ποδήλατό μου, τότε θα συναντήσω προβλήματα. Θα πρέπει να αλλάξω τρένο δύο έως τέσσερις φορές. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως ε, τις δυνατότητες που έχουμε. Παρότι η Ευρώπη επενδύει σε ε, σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλή ταχύτητα. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω, εσάς στην Επιτροπή Μεταφορών, να αλλάξετε την κατάσταση και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες αυτές και για τον τουρισμό. Σκεφτείτε την οικονομία του ταξιδιώτη όταν επενδύεται στις μεταφορές. Και όταν μιλάμε για τις μεταφορές δεν μιλάμε μόνο, μόνο για γραμμικές υποδομές όπως είναι οι σιδηροδρομικές γραμμές, μιλάμε και για διασυνοριακές υπηρεσίες, την έκδοση εισιτηρίων, την πληροφόρηση, την ε, προώθηση, την διαφήμιση δηλαδή, κάτι το οποίο είναι ε, ε, τομείς προβληματική. Να ενθαρρύνουμε τους τουρίστες να χρησιμοποιούν ε, βιώσιμες μορφές ενέργειας. Ε, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι ε, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα αεροπλάνα οι ταξιδιώτες, αλλά εάν θέλουμε να απαλλάξουμε από ανθρωπικές εκπομπές τις μεταφορές, θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτές τις πτυχές. Εξετάστε λοιπόν αυτά που ζητάμε. Ένα από τα πράγματα που ζητάμε είναι να συνεχίσετε να επενδύετε σε υποδομές μεταφορών, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ε, προοπτικές, τις δυνατότητες των ταξιδιωτών και ε, σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεχίσει να επενδύει σε τοπικές μεταφορές, σκεφτείτε για παράδειγμα τις θέσεις στάθμευσης για τα τουριστικά πούλμαν. Παρακαλώ, σκεφτείτε τις δυνατότητες των ποδηλατοδρόμων και για τους τουρίστες, όχι μόνο για την ε, απλή κινητικότητα. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και τις πολυτροπικές μεταφορές διότι το παράδειγμα που σας έδωσα αφορούσε ένα είδος μεταφορών. Εάν προσπαθήσει να συνδυάσει κανείς διαφόρους τρόπους μεταφορών, ε, απαιτείται η Ευρώπη να έχει καλύτερη στρατηγική και να ε, δει τα πράγματα από την πλευρά του ταξιδιώτη. Είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε ότι οι αερομεταφορές θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο και στο μέλλον. Θα θέλαμε όμως να σας καλέσουμε να εξετάσετε τον αντίκτυπο της, ε, πρωτοβουλία, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τον ενιαίο ουρανό, το Single Sky Initiative. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ο τομέας ε, του τουρισμού ε, στηρίζει τις προσπάθειές σας να προσελκύσετε περισσότερες επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών και θέλουμε να σας καλέσουμε να εξετάσετε τις δυνατότητες των ταξιδιωτών. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εμείς ως Επιτροπή είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Έτσι επιγράφει η Επιτροπή μας. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κριστίνα Νούνες από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για ένα εφόρο και ανταγωνιστικό τουρισμό. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη τιμή θα σας παρουσιάσω το μανιφέστο προτεραιοτήτων για την ε, αηφορία. Η πρώτη μας σύσταση εδώ θα ήταν ε, να δούμε την εγκάρσια διάσταση του τουρισμού, του αηφόρου και βιώσιμου κάθε φορά που γίνονται κάποιες δράσεις προγραμματισμού. Βεβαίως, ε, δεν είναι ένα θέμα μεμονωμένο, καλύπτει όλε τι πτυχέ του κλάδου και χρειάζεται την προσοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεύτερον, το Μανιφέστο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές για να ενθαρρύνει τον εθελοντικό έλεγχο για την προώθηση ε, του συστήματος ήτης που είναι για δείκτες τουρισμού, για τη βιώσιμη και αηφόρο διαχείριση ε, και εκτίμηση να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, οι προτιμήσεις και οι τάσεις ε, στον τουρισμό. Οι δείκτες αυτοί λοιπόν χρειάζονται και συντονισμό και συμβατότητα με ε, το παρατηρητήριο για τον εικονικό τουρισμό και τα δορυφορικά συστήματα. Θα πρέπει τα διάφορα μέσα που έχουμε να είναι συντονισμένα διαλειτουργικά από τη βάση προς την κορυφή και για διάφορους προορισμούς. Εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ποτέ αυτό που δεν μπορούμε να μετρούμε. Ε, και όλα αυτά ε, συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, με τη διαχείριση και για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε προσπάθεια και η σε οποιοδήποτε επίπεδο ε, διακυβέρνησης και διαχείρισης χρειάζεται μετρήσιμους συγκρίσιμους δείκτες για να μετρούμε και τις επιδόσεις. Ε, η βιωσιμότητα σημαίνει και οικονομική διάσταση και κοινωνική και γενικότερα ζητήματα που πρέπει να δοθούν ολοκληρωμένα. Και τέλος θα ζητούσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, και ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού ε, νόψη και της προσεχούς επαιτίου θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα για τον ανταγωνιστικό τουρισμό, το βιώσιμο, συστήματα, τεχνολογία και υποδομές. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι ο τουρισμός είναι κάτι που έχει να κάνει με συγκεκριμένο τόπο, χρειάζεται όραμα, μακροχρόνιο και προστασία των πόρων για να γίνουν όλα αυτά και όταν γίνουν θα συνεισφέρουν και προς την προστασία του κλίματος. Υπάρχει το θέμα της αηφορίας και της βιωσιμότητας και στον πολιτισμό ε, και το ζήτημα της ποιότητας ζωής, του τρόπου ζωής ενός τόπου ε, και εκεί θα πρέπει να συνεργαστούν διάφορες γενικές διευθύνσεις και θεσμικά όργανα καθώς επίσης και διεθνείς οργανισμοί με τελικό στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας η Κέρστεν Χόβαλτ ε, από τα Συνδικάτα των Εργαζομένων ε, στον κλάδο της Εστίας και της Γεωργίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε και κύριοι Ευρωβουλευτές, να σας παρουσιάσω τι ε, τις επίγουσες προτεραιότητές μας για τα προσόντα και τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε στον τουρισμό. Όπως ξέρετε, και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων καθόρισε τις ε, δεξιότητες, ε, την ε, κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση ως ουσιώδη στοιχεία, θεμελιώδη στοιχεία για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για την ισότητα ευκαιριών απασχόλησης. Θεωρούμε ότι στον τουριστικό τομέα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση, κατάρτιση όντω είναι προσαρμοσμένη στι ανάγκε των εργαζομένων και του κλάδου. Πρέπει λοιπόν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα ο τουρισμός, για παράδειγμα, πρόσβαση σε πληροφορική, θέματα ευαισθησιών και αλλεργιών ε, σε τρόφιμα. Ξέρουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες ε, στον ε, τουριστικό κλάδο είναι μικρομεσαίες, άρα χρειάζεται ειδική κατάρτιση του προσωπικού τους, γιατί πολύ συχνά οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να δώσουν μακροχρόνια άδεια στο προσωπικό τους για να καταρτιστούν. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες επιγραμμικής κατάρτισης. Αλλά δεν χρειάζεται να επανεπινοήσουμε τον τροχό. Πολλά γίνονται ήδη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες της Κομισιόν, ΕΜΠΛ, ΕΑΚ και Growth που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι η καλύτερη ε, επίβλεψη, καλύτερη χρηματοδότηση, καλύτερη ανταλλαγή ε, βελτίστων πρακτικών για την κατάρτιση και τις δεξιότητες. Να δούμε λοιπόν όλα τα δίκτυα, όλες τις προτάσεις που έχουν ήδη γίνει. Δεύτερον, ξέρουμε ότι στον τουρισμό ε, έχουμε πολλούς νέους εργαζόμενους. Για πολλούς είναι η πρώτη τους δουλειά. Είναι η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Άρα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά, ούτως ώστε ο τουρισμός να είναι ελκυστικός για τους νέους ως απασχόληση με βάση τα μέσα που ήδη έχουμε, την ε, εγγύηση για τους νέους, ε, τη συμμαχία για τις θέσεις μαθητείας, άλλες πρωτοβουλίες που έχει προτείνει η Επιτροπή σας και εδώ πρέπει βεβαίως να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αλλά πρέπει να έχουμε και νέα καινοτόμα προγράμματα στα πλαίσια της κατάρτισης. Για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εποχικών εργαζομένων, να δούμε πώς θα τους καταρτήσουμε όταν ακριβώς δεν εργάζονται λόγω της εποχικότητας. Ίσως δεν υπάρχει επαρκής γνώση των δυνατοτήτων που, υπάρχει, που υπάρχουν για να βρει κανείς δουλειά στον τουρισμό. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια δικτυακή πύλη για τον τουρισμό. Πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα το κάνουμε. Και επίσης το θέμα δεν είναι μόνο να προσελκύσουμε εργαζόμενους, αλλά να μείνουν και στον τουρισμό. Είμαστε όλοι πεισμένοι ότι πρέπει να κάνουμε πιο πολλά για να είναι καλές ε, θέσεις εργασίας, με ισότητα ευκαιριών, με αξιοπρεπή αμοιβή κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Και τώρα στο Λούις Δεγκράνδες Πασκουάλ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε και επτά οργανώσεις που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Το είπε και ο Πρόεδρος Κράμερ. Η Επιτροπή του Τιδό δεν είναι μόνο Επιτροπή Μεταφορών, είναι και τουρισμού. Και θα ήθελα να συγχαρώ εκείνους που εκπώνησαν το συγκεκριμένο μανιφέστο, γιατί συνδυάζει Ε, με έναν τρόπο πάρα πολύ ευφυή το πώς θα ξεπεράσουμε το άρθρο 197 της συνθήκης, 195 συγγνώμη. Ε, και κατά πόσο ε, θα δημιουργηθεί το πλαίσιο εκείνο για να προωθηθεί ο τουρισμός. Επανειλημμένα το έχουμε δει στο Κοινοβούλιο και θα το τονίσουμε. Το μανιφέστο συμπεριλαμβάνει όλα τα θετικά και τα απαριθμεί. Τι σημαίνει ο κλάδος του τουρισμού και ποια είναι η τεράστια κοινωνική διάσταση που είναι διπλή. Δημιουργεί θέσει εργασίας και επιτρέπει την ανταλλαγή ε, ανθρώπων ε, σε θέματα πολιτισμού. Είναι εγκάρσιος όμως ο χαρακτήρας, δεν εναρμονίζεται ε, προφανώς, αλλά με έμεσο τρόπο μπορεί να υπάρξει αποφασιστική επιρροή όλων των δραστηριοτήτων χώρες όπως η δική μου έχουν τον τουρισμό ως τον υπαριθμό ένα κλάδο της οικονομίας. Κάθε μέρα είναι μεγαλύτερος ο πλούτος και για τις αναδυόμενες ε, χώρες που ε, ψάχνουν έναν τρόπο να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, να αξιοποιήσουν ε, τις αρετές τους. Ευχαριστώ για το μανιφέστο. Είναι πάρα πολύ καλή ε, άσκηση. Ξεπερνάει τα προβλήματα της συνθήκης με έναν τρόπο πάρα πολύ λεπτό και ευφυή ε, να κινητοποιήσει εκείνα τα στοιχεία που πολλές φορές ε, τα έχουμε και εμείς αναφέρει, όπως είναι η εποχικότητα, αλλά έχουμε και ειδική εδώ. Το θέμα δεν είναι τώρα ε, ο τουρισμός να έχει άπαξ ε, μία στιγμή δόξα ας πούμε, ή ένα 15 λεπτό, αλλά να είναι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας ε, κάτι το σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η Κλάουντια Ταπαρδέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον τομέα του τουρισμού, διότι ε, είναι τομέας ε, που χαρακτηρίζεται από ενότητα και αυτό δείχνει πώς μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω όλα. Στο μανιφέστο συμπεριλαμβάνονται πολύ σημαντικά θέματα. Πρόκειται το μανιφέστο για την φωνή του ευρωπαϊκού τουρισμού, η οποία όμως ε, δεν γίνεται πάντα επαρκώς ακουστή. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να μπορεί να, κάνει περισσότερα, διότι ο ε, ευρωπαϊκός τουρισμός ε, κάνει πολλά για την ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, φέρνει κέρδος κλπ. Πιο σημαντικό είναι όμως ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν στηρίζουν επαρκώς τον τομέα αυτόν. Ελπίζω η σημερινή ημέρα να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα ε, για να έχουμε μια νέα τάση. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά τα θέματα, διότι πολύ από εμά συμμετέχουμε σε διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό. Επίσης, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις διάφορες ε, συζητήσεις που έχουμε μαζί της, ε, επίσημες και άτυπες, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Και άλλωστε, όπως υπόθηκε, είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε επαρκώς με το θέμα του τουρισμού και μάλιστα αναλυτικά. Ε, να εξετάσουμε τους διάφορους ε, επιμέρους τομείς που είναι σημαντικοί για τον τουρισμό. Επίσης, πιστεύω ότι ο τομέας του τουρισμού στην Ευρώπη έχει κάνει πολλά. Για παράδειγμα, είχαμε έτος τουρισμού ε, και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό ήταν δική μας πρωτοβουλία ε, και είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση. Επίσης, ε, το 2018 είναι έτος ε, πολιτιστικής κληρονομιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός και για να καταλάβει ότι δεν αρκεί απλά ένα έτος, χρειάζονται πολλές δράσεις ε, για να αναπτυχθεί περαιτέρω τομέας αυτές. Περιμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ένα σχέδιο δράσης. Έχουμε λάβει σχετική υπόσχεση. Το μανιφέστο αυτό αποτελεί σημαντικό μέσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχέδιο δράσης. Ε, ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι Ευρωβουλευτές να καταλάβουν ότι χρειάζεται μια στρατηγική ανάπτυξη για τον τομέα του τουρισμού. Και Τα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε μια απολύτως πεπαλαιωμένη τέτοια στρατηγική που δεν έχει λάβει υπόψη ε, τις τις ε, πρόσφατες εξελίξεις. Και Μία τελευταία παρατήρηση. Συνομιλώ με εκπροσώπους Υπουργείων, με εθνικές αρχές και όλοι όταν μιλούν για την επικουρικότητα στον τουρισμό επαναλαμβάνουν το ίδιο. Λένε ότι χωρίς ευρωπαϊκή υποστήριξη, χωρίς επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που δεν βλέπουμε στο σχέδιο Juncker, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει και ο τρόπος υποστήριξης των κρατών μελών για να έχουμε αναπτύξει του τουρισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εύαντ. Η κυρία Εύαντ, συγγνώμη. Και εγώ καλωσορίζω ιδιαίτερα αυτή την ε, εξέλιξη. Ορισμένοι είπαν πως είναι πρωτόγνωροι. Είναι πολύ θαρρυντικό όλοι αυτοί οι φορεί να συνεργάζονται και να παρουσιάζουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και να θέτουν τον τουρισμό ως βασικό πολιτικό θέμα, όπως ε, πολύ καιρό επιχειρούμε να κάνουμε και εμείς. Πιστεύω λοιπόν ότι τα θέματα που καλύπτουν οι διάφορες παρουσιάσεις είναι ακριβώς απόδειξη του πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός, από πόσες πλευρές για τη ζωή μας. Βεβαίως, σωστή εστίαση στις μικρομεσαίες, πολύ σημαντικές για την οικονομία, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στον τουρισμό, όχι μόνο για το ταξίδι, τη μετακίνηση μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, αλλά και προσβασιμότητα για παράδειγμα. Πάντα το έχουμε τονίσει αυτό για τα άτομα με αναπηρίες. Και επίσης, βεβαίως ε, τονίζουμε ιδιαίτερα και την βιωσιμότητα, θα μπορούσαμε να τονίσουμε περισσότερο το ρόλο του τουρισμού ε, για να αντιμετωπιστούν ε, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, γιατί και αυτό είναι βασικό για τη δουλειά μας στο Κοινοβούλιο. Αλλά μια συγκεκριμένη ερώτηση για τις δεξιότητες και την κατάρτιση. Το μανιφέστο σας λέει ότι 25 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Ευρώπη βασίζονται σε συγκεκριμένες δεξιότητες ε, και πρακτικές ε, δυνατότητες που έχουν. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του, της Ουαλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και η στρατηγική μας ε, για τον τουρισμό στην Ουαλία λέει ότι δεν θεωρείται ποιοτική η απασχόληση στον τουρισμό. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και έχουμε μια οργάνωση που λέγεται πρώτα οι εργαζόμενοι και είναι οργάνωση επαγγελματικής κατάρτισης και λέει ότι έχουμε πολλά κενά σε ανθρώπους με συγκεκριμένα προσόντα και 25% των ε, εργοδοτών είπαν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό με τα προσόντα που χρειάζονται. Και σε σχέση με αυτό, βέβαια, υπάρχει το πρόβλημα του πόσο μπορούν να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Και το ανέφερε και κάποιος για τους νέους εργαζόμενους. ο αριθμός των νέων κάτω των 24 ετών που προσλαμβάνονται στον τουρισμό είναι τριπλάσιος από αυτόν που προσλαμβάνονται σε όλους τους άλλους τομείς. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός, να ενημερωθεί η κοινή γνώμη γενικά επ' αυτού. Πώς νομίζετε λοιπόν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής έμφαση στη σημασία του τουρισμού και στην αξία των προσόντων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Δείτε Κλούντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω. Το έγγραφο πραγματικά καλύπτει όλους τους ε, τομείς, εν συντομία, αλλά όλους τους σημαντικούς τομείς. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί. Να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Εύανς κατά προσόντα και την ανάγκη να προωθηθεί ο τουρισμός και ως κλάδος για σταδιοδρομία, γιατί δεν έχει δοθεί νομίζω επαρκής έμφαση εκεί και ε, στα catering υπάρχει πρόβλημα δεξιοτήτων και ε, προσόντων ε, γλωσσομάθειας. Γενικότερα στη φιλοξενία υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση των θέσεων εργασία και των δεξιοτήτων. Και δεν είναι γενικώ κάποια προσόντα, είναι μια ολόκληρη σειρά συγκεκριμένων προσόντων και η Ένωση Ξενοδόχων θεωρεί ότι είναι πρώτη προτεραιότητα και έχει να κάνει και με την εκπαίδευση. Και θα πρέπει να προωθείται ε, και αυτός ο κλάδος, να σκέφτεται δηλαδή, κανείς να σταδιοδρομήσει και στον τουρισμό. Ευχαριστώ, Γιάννη Σνίλς. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι επικροτώ το μανιφέστο αυτό. Νομίζω ότι θα αποτελέσει χρήσιμη βάση για τη συνέχιση των εργασιών που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα. Θα αναφερθώ πρώτα στην δική μου περιφέρεια και κατόπιν θα υποβάλω δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις προτάσεις. Προέρχομαι από την Βόρεια Σουηδία, από περιοχή που κατά τη διάρκεια της ε, δεκαετίας του 90 αποφάσισε ότι ο τουρισμός ε, θα είναι η βάση της ε, οικονομίας μας. Ε, χρησιμοποιήθηκε το, ε, χρησιμοποιήθηκαν τα διαφορετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε κατανομή των πόρων για να γίνουν επενδύσεις. Έχουμε δώσει σημασία στη βιωσιμότητα. Έχουμε συνδέσει την ε, τοπική κουζίνα με τον τουρισμό. Και είδαμε θετική ε, ανάπτυξη όλης της περιφέρειας. Εφόσον είμαστε εμείς αρμόδιοι για τον τουρισμό και η Ρέγγι είναι ε, αρμόδια για την περιφερειακή ανάπτυξη θα πρέπει να συνεργαστούμε στο θέμα του τουρισμού, όπως ε, και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι τοπικές δράσεις για τον τουρισμό. Εκεί δημιουργούνται οι θέσεις απασχόλησης, εκεί υπάρχει ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Χρειάζεται φυσικά και προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη σήμερα χρησιμοποιούνται πολλοί πόροι από τα διευθυντικά ταμεία για την ανάπτυξη του ε, τουρισμού δύο προτάσεις. Να εκπονηθεί μελέτη μαζί με την Επιτροπή ΔΕΕΚΙ, να δούμε τι ενισχύσεις δίδονται στον τουρισμό στα διαρθρωτικά ταμεία. Εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά ίσως το ξέρει η Επιτροπή ΔΕΕΚΙ, ίσως το ξέρει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η άλλη μου πρόταση είναι να επιλέξουμε 10-15 περιφέρειες της Ευρώπης που έχουν αποφασίσει ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό ταμέα της οικονομίας. Υπάρχουν και άλλες περιφέρειες της Ευρώπης, πέρα από τη δική μου που το έχουν αποφασίσει αυτό. Και ας μάθουμε η μία περιφέρεια από την άλλη. Και να ε, ενσωματώσουμε ε, τους ε, βασικούς στόχους της περιφέρειας αυτής στην τουριστική στρατηγική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κλάουτια Μοντέρα Δακλήρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα σύντομα, χωρίς να επεκταθώ γιατί εδώ είναι όντως Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Και κάτι που βλέπουμε και είναι ξεκάθαρο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές μας ή την ιδεολογία μας, ε, συμφωνούμε όλοι για τον τουρισμό και με το συγκεκριμένο μανιφέστο δίνεται ευκαιρία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα να προχωρήσουν σε ένα κοινό στόχο και να αποδείξουν ότι ακριβώς αυτός ο οριζόντιος εγκάσιος χαρακτήρας του τουρισμού έχει κοινά στοιχεία που πρέπει να αξιοποιούνται. Αυτό το βλέπουμε παντού σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σε όλα τα πολιτικά μέτωπα. Είναι πολύ θετικό το μανιφέστο και εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια. Διότι ορισμένα από τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο μανιφέστο μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόοδο ε, της οικονομίας. Ακούστηκαν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός αλλά μπορούμε με μεγάλη ικανοποίηση να διαπιστώνουμε ότι πολλές από τις προτάσεις μας συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο μανιφέστο. Χαίρομαι λοιπόν που ε, ομονοούμε τόσο πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι ο στόχος είναι κοινό να αναπτυχθεί ο τομέας και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Τα θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχής γενομένης από το Κοινοβούλιο και από τούτο την Επιτροπή, αλλά και μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αγωνιστούμε για να αυξηθεί ο τουρισμός, να ενισχυθεί η στήριξή του. Πραγματικά δημιουργεί θέσεις εργασίας και απασχόληση παντού. Δεν θα πρέπει να αφιστούμε κόπων και προσπαθειών, να συνεχίσουμε με μία φωνή να υπερασπιζόμαστε τον τουρισμό. Είπαν και άλλοι συνάδελφοι ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό το μανιφέστο, είναι πολύτιμο και είναι όμως μια αφετηρία και μόνο. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να προχωρούμε στη σωστή κατεύθυνση. και το πρόγραμμα δράση αυτό να γίνει πραγματικότητα. Χρηματοδότηση, βέλτιστες πρακτικέ, όλα αυτά είναι στοιχεία πολύ χρήσιμα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πάντα σεβόμενοι την αρχή της επικουρικότητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Θα πρέπει όμως να αναζητούμε πάντα κοινού στόχους για να συνεργαζόμαστε και να ε, πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο σημαντικό είναι αυτό ο κλάδο για τι οικονομίε των χωρών μα. Και επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ γιατί τα θέματα δεν είναι μονοσήμαντα. Δράτω με τις ευκαιρίες που αριβρίσκεται εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, κάνω μερικά ερωτήματα. Το έγγραφο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το μανιφέστο αυτό, και είναι και πολύ καλά ε, πώς να το πω, προετοιμασμένο. Ήταν πολύ καλή η διαδικασία εκπόνησης. Όλα αυτά είναι ωραία. Πώς μπορούμε αυτά που συζητούμε εμείς εδώ να τα μεταφέρουμε ε, επιτόπου. Η Επίτροπος ε, μίλησε για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. Πώς θα γίνει αυτό. Ερωτώ, πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να τα μεταφέρουμε αυτά στον κόσμο και να μην έχουμε επικαλύψεις. Θα ε, πρέπει να εκφράσω και ένα παράπονο τώρα. Είχα κάνει μια πρόταση στο παρελθόν γιατί θέλαμε το έγγραφο αυτό να φτάσει μέχρι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν θέλουμε αυτά που μας απασχολούν εμάς να φτάνουν και στους ενδιαφερόμενους και σε όλους τους φορείς του τουρισμού, πρέπει αυτοί να ενημερώνονται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μαθαίνουν τι συμβαίνει. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν στην πρόσβαση. Μπορεί να μεταφραστεί το μανιφέστο ε, οδηγός αυτός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να έχουν πρόσβαση όλοι αυτοί οι φορείς του κλάδου. Δεν ξέρω αν θα το μεταφράσετε. Κάποτε άκουσα ότι θα γίνει αλλά υπάρχουν κάποιες γλώσσες που εξαιρέθηκαν, όπως είναι το πορτογαλικά. Ε, τι θα γίνει, αυτό είναι εμπόδιο. Αυτή είναι η μικρή δυσφορία όμως, με το παράπονο που θα ήθελα να σας αναφέρω. Ας έχει όμως. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε διάφορες πλατφόρμες, μελέτες, μανιφέστα, πολύ σημαντικά και κρίσιμα. Θα πρέπει να φτάνουν πάντα στα χέρια των ενδιαφερομένων. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει και να τα αντιμετωπίσουμε. Και όλοι έχουμε κοινό συμφέρον ε, να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Η Επιτροπή μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο μεταφορών, είναι και τουρισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ιζαβέλα Ντεμόντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας που μας παρουσίασαν ε, την κατάσταση. Είναι η μόνιμοι συνομιλητές μας ε, και είναι οι θεμελιώδεις ε, φορείς που εργάζονται και θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε την πολιτική μας. Και αυτή σίγουρα είναι η σωστή προσέγγιση. Ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι θέμα μόνο διαχείρισης ε, από το δημόσιο τομέα και ο ιδιωτικό τομέας πρέπει να παίξει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Και παραλαμβάνω, είναι ένα ολόκληρο είναι ένας ολόκληρος κλάδος. Ο τουρισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο απλώς ε, ένας πάροχος υπηρεσιών. Είναι ένας συνολικός κλάδος οικονομίας και πρέπει να θεωρηθεί ως κλάδος και είναι ο τρίτος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να στηριχθεί με όλη την αναγκαία αφοσίωση και αποφασιστικότητα. Και κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ό,τι επενδύεται στον τουρισμό είναι κάτι το οποίο ωφελεί και τις περιοχές μας, ε, ωφελεί το τοπίο. Οφελεί, ε, για παράδειγμα, την ελκυστικότητα ε, ε, μιας περιοχής. Αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών σε αυτή την περιοχή. Είναι λοιπόν ένας κλάδος για τον οποίο η Ένωση πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια. Πρέπει πραγματικά να είναι αιστεία για τις επενδύσεις μας, γιατί υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τον τουρισμό στην Ευρώπη, βεβαίως. Και υπογραμμίστηκε και αυτό. Και υπάρχει και το θέμα της φορολογικής πολιτικής. Πρέπει να το μελετήσουμε αυτό. Πρέπει να είναι ε, παρόμοια η φορολόγηση για να υπάρχει θεμητό ανταγωνισμό. Γιατί αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και να προσθέσω και κάτι άλλο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ συγκεκριμένα και απτά. Υπάρχουν ε, τοπικοί φόροι, για παράδειγμα φόροι επί των διανυκτερεύσεων. Δεν έχω από πλευρά αρχή αντίρρηση, αλλά πρέπει να υπάρχουν προποθέσει. Στην πόλη μου, για παράδειγμα, ο φόρο επί των ε, διανυκτερεύσεων ξεκινάει από 4,5 ευρώ και μπορεί να πάει και πολύ παραπάνω. Δεν νομίζω ότι αιτιολογείται κάτι τέτοιο. Πρέπει... Τι έννοια έχουν αυτοί οι φόροι. Οι φόροι επί των διανεκτερεύσεων πρέπει να δεσμεύεται αυτός που τους συλλέγει ότι θα επενδυθούν μετά στον ίδιο τομέα. Τώρα, κάτι άλλο, το θέμα της ψηφιοποίησης. φυσικά ψηφιοποίηση ε, δεν σημαίνει μόνο η έρευνα που κάνουν οι καταναλωτές στο web. Το θέμα είναι να υπάρχουν επαρκή στοιχεία όταν κάποιος κάνει μια, ε, ένα search, μια έρευνα ε, στο ίντερνετ. Και κάτι άλλο επίσης που είναι ίσως ο αδύναμος κρίκος. Είναι οι αστικές μεταφορές στους χώρους όπου μεταβαίνουν οι τουρίστες δεν αξιοποιούνται αρκετά, δεν είναι αρκετά γνωστές οι δυνατότητες τοπικών μεταφορών και πρέπει να υπάρχει ε, και ε, ε, μια διεύρυνση του δικτύου, να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια. Μόνο με αυτές τις μορφές τουρισμού, συγγνώμη, μεταφορών, που βέβαια πρέπει να είναι συμβατές με το περιβάλλον, μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τους καταναλωτές, τους τουρίστες. Είναι σημαντικό να υπάρξει ε, δράση σε όλα τα επίπεδα. Είναι απόλυτα θεμελιώδες αυτό για αυτό το τόσο θεμελιώδη για την απασχόληση τομέα της οικονομίας μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της εργασίας. Μια μικρή μόνο παρατήρηση. Ακούσατε όλους τους βουλευτές να μιλούν με διαφορετικό τρόπο και εκπλήσωμαι πάρα πολύ. Ε, μιλήσαν 7-8 εκπρόσωποι και ο πρόεδρος ε, από εσά και μιλήσαν όλοι αγγλικά. Εμείς μιλάμε καθένα στη γλώσσα του. Η Ευρώπη έχει ένα πλούτο, μια παράδοση και ο τουρισμός περνάει από όλα αυτά. Και αν δεν τα σεβόμαστε δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό. Ε, εγώ είμαι από τη Γαλλία, που είναι η πρώτη χώρα σε τουρισμό στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι η πρώτη σε τουρισμό στον κόσμο. Και είμαι αντιπεριφερειάρχης στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ευρώπης, Provence Alpes Côte d'Azur, που μετά το Παρίσι είναι και ο πρώτος ε, προορισμός. Και είμαι αυτοδιοικητικός ερετός και βλέπω ο καθένας να κάνει προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρχει παντού ο, τουρισμός με διαφορετική προσφορά και δεν πρόκειται η Ευρώπη να τα υλοποιήσει όλα αυτά. Τι διαπιστώνω τώρα. Εγώ είμαι από τη Μασαλία. Ε, είχαμε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Θεωρείται μεγάλη πολιτιστική πόλη η Μασαλία, ωστόσο αυτό που έγινε ε, μας επέτρεψε να έχουμε στόχο 12 εκατομμύρια τουρίστες και ήρθαν 14. 2 εκατομμύρια το χρόνο έκτοτε. Όταν έχεις ένα σήμα ε, μια τεχνογνωσία που σου αναγνωρίζεται, γίνονται τα πράγματα. Και τα πράγματα μπορεί να γίνονται τεχνικά με το Wi-Fi, με τρένα, ποδήλατα, αεροπλάνα και βαπόρια και κατάρτιση. Ε, κάθε περιφέρεια με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητές της και τις αρμοδιότητες κάνει την προσφορά της. Και έτσι ολοκληρωνόμαστε. Προφανώς είναι πολύ μεγάλος και έντονος ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και υπάρχει ε, ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε είναι η τρομοκρατία ε, και οι επιθέσεις. Στην Ιορδανία υπάρχει η Πέτρα. Ποιος πάει στην Πέτρα σήμερα τουρισμό και είναι οι Ιορδανοί καταπληκτικοί άνθρωποι. Στην Τινησία δεν πατάει η ψυχή ε, γιατί ο κόσμος φοβάται. Δεν έχουν αλλάξει την ίση, είναι εξίσου θαυμάσιοι άνθρωποι. Στο Παρίσι είδαμε ότι μειώθηκε κατά 20% η κίνηση και ο τουρισμός μετά τις επιθέσεις. Όλα αυτά είναι μεταβατικά μέχρι να τα ξεχάσει ο κόσμος που τα ξεχνάει και γρήγορα από ό,τι μαθαίνουμε. Ε, αλλά στην Ευρώπη εμείς, σε αντίθεση με την Αφρική, την Νότια Αμερική, ε, δεν έχουμε μόνιμη κίνηση. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Ακαπούλκο. Ε, στο Ακαπούλκο θυμάστε που πήγαινε ο κόσμος και βουτούσε από τους βράχους τώρα δεν τολμάει να πατήσει στο Ακαπούλκο γιατί το τον δολοφονούν. Στην Ευρώπη δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στην Αφρική, στην Νότια Αμερική βίας. Ε, άρα ε, και το λέω προς τους συναδέλφους και δεν χωρέ εδώ δεξιά και αριστερά. Ο τουρισμός ε, υπερασπίζεται τους τόπους μας με βάση την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα ή την Ευρωπαϊκή Αθλητική Πρωτεύουσα ή την Ευρωπαϊκή Τουριστική Πρωτεύουσα. Θα μπορούσαμε κάθε χρόνο να έχουμε άλλη χώρα, άλλο θέμα, όπως είναι οι παράκτητες περιοχές, η θάλασσα, η εξοχή, η βιοπικιλότητα, το βουνό ή ακόμα και ε, διάφορες ε, τουριστικές διαδρομές, γαστρονομικό τουρισμό. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων. 5, 6, 7, 8, 10 πόλεις ε, θα έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτό και θα αξιοποιεί τον τουρισμό, ε, το, το folklore, ξέρω εγώ, στη Σουηδία, τα το, ε, τοπία στην Πορτογαλία, την Κανμπιέρ, την περίφημη λεωφόρο στη Μασσαλία κτλ. Ή, ή την ποιότητα ζωής στη Μασσαλία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κύρκος, παρακαλώ. Thank you, Chair. Θα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το μανιφέστο το οποίο μας παρουσιάστηκε σήμερα και ε, η συνεργασία των εκπροσώπων ε, των φορέων του ταξιδιού και του τουρισμού και η έκκληση που κάνουν στα ευρωπαϊκά institutions ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και την Ευρώπη να παραμείνει ελκυστικός προορισμός αλλά και κυρίως η ευρωπαϊκή βιομηχανία του τουρισμού να παράξει περισσότερε θέσει εργασία. Ειδικά για χώρε που βρίσκονται στην κρίση, όπω η δική μου αλλά και άλλε, βλέπουμε πω ε, ο τουρισμό σε αυτέ τι περιπτώσει αποτελεί ίσω τον ε, κυρίαρχο τομέα που δημιουργούνται νέε θέσει εργασία. Και μια και μίλησα και για την κρίση, να σα ε, μεταφέρω και την επίσκεψη του Δημάρχου Λέσβου στη Λίμπε την προηγούμενη εβδομάδα όταν μιλάμε για κρίση φαντάζεστε ένα νησί με 400.000 διελεύσεις προσφύγων και μεταναστών το νησί έχει 30.000 κατοίκους και όμως ο Δήμαρχος μας εξήγησε και μας απέδειξε ότι ε, η παρουσία τόσων ανθρώπων εκτός από τις πρώτες μέρες έγινε σε κέντρα φιλοξενίας με πολύ καλές συνθήκες και το νησί αυτή τη στιγμή αποτελεί έναν προορισμό για χιλιάδες τουρίστες. Φοβόντουσαν πτώση 80% και το νησί είναι κλεισμένο ε, για πολλούς μήνες. Αυτό δείχνει ότι αυτό που εύκολα λέμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές αξίες, οι πολίτες της Ευρώπης το αποδεικνύουν με τον δύσκολο τρόπο που είναι πληρώνοντας για να πάνε στο νησί της Λέσβου και ξοδεύουν τις λίγες διακοπές τους για να δούνε ένα νησί το οποίο υποδέχτηκε τόσες χιλιάδες πρόσφυγες χωρίς να ε, καταρρεύσει η τοπική κοινωνία. Αντί θα τους αγκάλιασε με τον καλύτερο τρόπο. Ε, βλέπουμε λοιπόν όταν μιλάμε για Ευρώπη ε, καινούριο Ευρώπη ισχυρό προορισμό τουριστικό υπάρχουν πάρα πολλέ πλευρές που δεν έχουμε ακόμα εξετάσει και είναι πολύ σημαντικό να τις εξετάσουμε και αυτές. Δύο πράγματα θα κρατήσω από το μανιφέστο, όλα είναι ενδιαφέροντα αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο. Το ένα είναι η συνεργατική οικονομία και η επέκταση των υπάρχοντων νόμων ή η δημιουργία ενό νέου πλαισίου. Στην Ελλάδα είχαμε 15% αύξηση των αφήξεων του τελευταίου μήνε με 3% μείωση των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία. Αυτό το 18% που εξαφανίστηκε ξαφνικά από το ραντάρ προφανώ πήγε σε μια οικονομία η οποία δεν υπάρχει, για την, ε, για τον, δεν προσφέρει στην εφορία, δεν προσφέρει στην οικονομία μα, απλώ υπάρχει και καταναλώνει τις, ε, τους, τους πόρους. Και το δεύτερο είναι η πολύ σωστή διαφάνεια και ουδετερότητα για τις ε, έρευνες στο ίντερνετ και όχι μόνο μουσική, αλλά και οι μαρτυρίες των ε, επισκεπτών πρέπει να εξασφαλίζεται πως είναι σε ένα καθεστώς διαφάνειας και αξιοπιστίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον πως το ραπόρ Del Monte, το Monte, το οποίο βγάλαμε το Σεπτέμβριο, αναλύει αυτά ακριβώς τα θέματα σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος και εδώ δημιουργείται και μία απορία πώς από αυτό το ρεπόρτ, το οποίο πραγματικά είναι η έκφραση του Κοινοβουλίου πάνω στα θέματα του τουρισμού, πώς θα μπορούμε να πάμε στα επόμενα βήματα που είναι η διερεύνηση σε κάθε κλάδο και σε κάθε τομέα, πώς μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα που περιέχονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο τώρα στους ομιλητές μας, να κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Ο Άνταμ Μπόντο αναφέρθηκε στον τρόπο έκδοση των εισιτηρίων, το Κοινοβούλιο, ήδη αποφάσισε πριν από 8 χρόνια με το Συμβούλιο, στο τρίτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους, ότι τα εισιτήρια πρέπει να περιέχουν όλες τις προφορίες παντού στην Ευρώπη. Και είπαμε ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να μπουν όλοι σε όλα τα τρένα, ακόμη και τα υψηλή ταχύτητα, αλλά ε, δυστυχώς το Συμβούλιο το αποδυνάμωσε αυτό. Γιατί είπαν ότι στο μέτρο που δεν, δεν ε, δυσχεραίνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Πρέπει όμως οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να ασκήσουν επαρκή πίεση στην, Αυστρία. Ξέρω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι δυνατόν να, συγγνώμη, να, θα είναι δυνατόν να πάρει και το ποδήλατο του. Για το ποδήλατο αναφερόμουν προηγουμένω. Το ποδήλατο να μπορεί να μπει σε όλα τα τρένα. Είπαμε λοιπόν ο τουρισμός ε, ε, έχει τεράστιες ε, θετικές επιπτώσεις στο εισόδημα ακόμη μεγαλύτερο και από τις κρουαζιέρες και οι κρουαζιέρες βέβαια είναι πολύ καλές αλλά Πολλέ φορέ στη Βενετία, για παράδειγμα, λένε ότι δεν μπορούν πια να δεχθούν τόσο μεγάλα κρουαζιερόπλαια, δημιουργούν προβλήματα. Άρα πρέπει να τα δούμε αυτά τα προβλήματα από του επισκέπτε. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να απαντήσετε ε, με τη σειρά που πήρατε και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας ε, απαντήσουμε γραπτός σε όλες τις ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και τα καλά σας λόγια. Θα θέλαμε όμως υποστήριξη στην πράξη. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με το να υπάρχει μια ε, εξωτερική μονάδα για τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι επαρκής ο προϋπολογισμός για τον τρίτο μεγαλύτερο οικονομικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, υποστηριχθεί περισσότερο ο τουρισμός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και την ε, ομάδα του κύριου Κοράτσα, διότι χρειάζονται περισσότερους πόρους και περισσότερη υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Θα συνεχίσω στα γαλλικά για τον Γάλλο συνάδελφο. Εγώ σπούδασα στο Έξαν Προβάνς, αλλά πάνε χρόνια. Ε, ζητώ συγγνώμη που ήταν όλα στα αγγλικά. The reason why it was in English is because... Ε, μίλησα στα αγγλικά γιατί... Ε, ε είναι άτυπο ο τρόπος με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Χρήματα δεν είχαμε και πόρους, γι' αυτό ήταν υποχρεωτική η εργασία μας στα αγγλικά. βεβαίω για να πιάσει τόπο θα πρέπει να μεταφραστεί το μανιφέστο και δεν θα πρέπει να είναι μόνο μια βάση για εργασία στις Βρυξέλλες, προφανώς. Εκεί μπορούν οι ευρωβουλευτέ να διαδραματίσουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Να το μεταφέρετε τις δικές σας περιφέρειες, να δούμε τι χρειάζεται και ε, τι ανάγκες υπάρχουν και μια σύνοψη στις κατοτόπους γλώσσες θα μας βοηθούσε για να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τα μελήματα που πολύ σωστά αναφέρατε. Ευχαριστώ. Ο Χριστιαν συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφο. Συμφωνώ. Βεβαίω έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία και σκεφτόμαστε και το δυναμικό τώρα. 100 εκατομμύρια τουρίστε θα μπορούσαμε τα επόμενα 15 χρόνια να έχουμε επιπλέον στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται μια κοινή στρατηγική που να σέβεται ε, τους, ε, ε, διαφόρους φορείς επιτόπου. Έχουμε τη δυνατότητα, αλλά χρειάζεται και μια στρατηγική για να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να έρθουν 100 εκατομμύρια τουρίστες. Βεβαίως, ε, η κατάρτιση είναι στον πυρήνα της στρατηγικής μας και είναι η κεντρική ιδέα για να έρθουν αυτοί οι νέοι ε, πελάτες και νέοι και ικανοποιημένοι. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον σας, για τη σκληρή δουλειά σας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία καθημερινά συνεργαζόμαστε. Ε, Βεβαίω χρειάζεται και τη δική σας υποστήριξη και περισσότερα κονδύλια για να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει αυτή η νέα στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο Άνταμ Μπόντορ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Νίλσον σχετικά με την χρηματοδότηση. Όταν μιλάμε για χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον τουρισμό, μιλάμε για ένα ή δύο εκατομμύρια ευρώ που ε, διατίθενται αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι αγωνίζεστε να αποκτήσετε περισσότερους πόρους για τις μεταφορές. Ε, μιλάτε όμως για δισεκατομμύρια και τώρα μιλάμε για λίγα εκατομμύρια στα οποία γίνονται και όλες περικοπές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο δεν ενθάρρυνε τις περιφέρειες να επενδύσουν στον τουρισμό. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει ο τουρισμός να παίξει συγκεκριμένο ρόλο και θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και να τα βοηθήσουμε να επενδύσουν στον τουρισμό. Ε, ευχαριστώ, κύριε Νούνες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, Μία τελευταία παρατήρηση για την βιωσιμότητα και την ε, ανταγωνιστικότητα. Ε, την καταπολέμηση των εποχιακών διακυμάνσεων, να παρατείνουμε δηλαδή τις τουριστικές εποχές, είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορούμε, το οποίο δεν μπορούμε να καλύψουμε σήμερα. Θα συμπεριλαμβάνεται όμως τις γραπτές μας απαντήσεις. Και ο όρος κλειδί για μας είναι ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την προστασία του τουρισμού και όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι υπάρχει ανάγκη για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ε, περιφερειών ε, που έχουν ε, θέση στο κέντρο της οικονομικής ζωής τον τουρισμό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Πολύ ευχαριστώ θα συνεχίσουμε όμως και χρειαζόμαστε υποστήριξη διότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες που μας λείπουν. Ε, υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη, χρειαζόμαστε όμως περισσότερα στοιχεία. Επίσης θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω για την ε, υποστήριξή σας προς την πρωτοβουλία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Κέρστιν Χόβαλτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Τζι Evans ε, και ε, την ε, συνάδελφο που μίλησε για την κατάρτιση, τα προσόντα και τις δεξιότητες. Παραμένουν τα προβλήματα και ε, πραγματικά αυτό που χρειάζεται είναι συντονισμένη δράση. Θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν. Οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρμόδιε γενικέ διευθύνσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι παντού στου διάφορου κλάδου του τουρισμού. Χρειάζεται οπωσδήποτε συνεργασία. Είναι πολλά τα μέσα, τα εργαλεία, οι πρωτοβουλίε, τα project πρέπει να συντονιστούν για να αποδώσουν. Οι κοινωνικοί εταίροι Ακούσαμε τι κάνουν ε, το μέσο της εστίασης ε, ε, με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη μαθητεία να γίνει πραγματικά μια ποιοτική μαθητεία. Στη φιλοξενία έχουμε προγράμματα, έχουμε ταχύ ρύθμα, τμήματα εκπαίδευσης, προσφύγων για να έρχουν γρήγορα στην αγορά εργασίας. Είναι μια σειρά τα ζητήματα και οι πρωτοβουλίες που μπορούμε να βασιστούμε και να προχωρήσουμε και να οικοδομήσουμε σε αυτά. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Μπορεί να γνωρίζετε ότι η βάση του τουρισμού να έχει ο κόσμος το χρόνο και τα χρήματα για να κάνει τουρισμό. Και φέτος το 2016 είναι η 80η επέτειος της σύμβασης του ILO που εγκρίθηκε το 26 για ε, πληρωμένες διακοπές. Πριν από 80 χρόνια, πότε ήταν. Ε, το 36 προφανώς. Και εμείς ε, από πλευρά συνδικάτων ε, θα το γιορτάσουμε στις 24 Ιουνίου στην ΑΚΕ και θα σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε αυτή την επέτειο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και τώρα και η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί. Είναι ο κύριος Κάρλο Κοράτσα, εκπρόσωπος της Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο γενικά για τη στήριξη και την ενθάρρυνση που δίνεται καθημερινά στην Επιτροπή για να ε, αναλάβει και νέες πρωτοβουλίες σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα και χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό αυτό το μανιφέστο να διευκολύνει πολύ τη δουλειά μας. Μας επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον κλάδο και διαπιστώνουμε ότι πολλές από αυτές είναι και στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επ' αυτών ε, κάνουμε και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Όπως τα ξέρετε, στις 5 Απριλίου είχαμε μία εκδήλωση με την παρουσία και του κυρίου Κράμερ σε πολύ ψηλό επίπεδο, με τη συμμετοχή και πολλών άλλων ευρωβουλευτών και τριών επιτρόπων. Όχι μόνο ο αρμόδιος επίτροπος, η αρμόδια επίτροπος η κυρία Νενκόφσκα, αλλά και ο επίτροπος που είναι αρμόδιος για την απασχόληση. Και εδώ είναι η επίτροπος η κυρία Ντίσεν και, ο Επίτροπος, και η Επίτροπος Κρέτου για τα περιφερειακά θέματα. Είναι νομίζω αυτό ένα σημαντικό μήνυμα ότι η Κομισιόν έχει μια εγκάρσια προσέγγιση. Συνεργάζονται διάφορες υπηρεσίε και έχει πλήρη συνέστηση της σημασίας για την ανάπτυξη και για την απασχόληση του τουρισμού. Σημερίζεται λοιπόν όλα όσα υπόθηκαν ο τουρισμός είναι κατά πάση πιθανότητα από τον οποίο μπορούμε να προσβλέπουμε σε περισσότερα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους και ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ε, ποσοστά ανεργίας 50% για τους νέους. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, συμφωνούμε. Η Επιτροπή πρέπει να κάνει περισσότερα με τους περιορισμένους πόρους που έχει. Πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους και τις πιστώσεις όλους ε, τους πόρους ε, του προϋπολογισμού, όχι μόνο κάποιων ε, προγραμμάτων. Και αυτή είναι η λογική και του προγράμματος Juncker. Δεν είναι μόνο για στρατηγικές επενδύσεις, είναι και καλύτερη εξοπλίση των υπαρχόντων των πόρων του προϋπολογισμού. Για να γίνει αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών από τις περιφέρειες, γιατί οι περιφέρειες αποφασίζουν τελικά για τη δαπάνηση ενός σημαντικού τμήματος του προπολισμού και πιστεύω ότι το μήνυμα που ήθελε να δώσει η Επίτροπος ε, η υπεύθυνη για τα περιφερειακά είναι ότι η περιφερειακή πολιτική πρέπει να βοηθήσει τον τουρισμό να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Και το ίδιο μήνυμα έδωσε και η κυρία Τίσεν. η ε, κοινωνική πόροι, οι εγγυήσει ε, για το πρόγραμμα για τους νέους, ο έρασμος συν, όλα αυτά πρέπει να συμβάλλουν ούτω ώστε η ανάγκη που έχει ο κλάδο για περισσότερου προσοντούχου να μπορέσει να καλυφθεί. Και επ' αυτού μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε πολύ συγκεκριμένε προσπάθειε. Στον προπολογισμό του COSME 2017 θα υπάρξει μια πίστοση 1 εκατομμύριο γι' αυτό. Και η Ντέζο Απασχόληση, ΕΜΠΛ, έχει θέσει τον τουρισμό ω ε, προτεραιότητα για την κατάρτιση. Θα μπορέσουμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε άλλα 3 εκατομμύρια γι' αυτά και βασιζόμαστε πολύ και στη συνεργασία με τον ίδιο τον κλάδο. Αυτή η εργασία για την κατάρτιση πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου. Θεωρώ ότι αν υπάρξει και περισσότερη κινητικότητα σε αυτά τα στάζου κατάρτισης, περισσότερη κινητικότητα μεταξύ βορρά και νότου, διότι ξέρετε ότι στην αγορά αυτή είναι πολύ μεγάλη η εποχικότητα. Νομίζω ότι έτσι θα βοηθούσαμε συγκεκριμένα τους νέους που ψάχνουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης για δουλειά. Για την συμμετοχική οικονομία. Όπως συζητείται η Επίτροπος Γενικόφσκα ανήγγειλε ήδη τις κατευθυντήρες γραμμές που θα υποβληθούν τον Ιανουάριο και σε αυτή τη φάση εκπονούμε μελέτες μαζί με τον κλάδο. Έχουμε συνέστηση ότι υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όχι μόνο πρόβλημα της ελευθερίας του επιχειρήν, αλλά είναι και πρόβλημα και ισοτήμων συνθήκων ανταγωνισμού που πρέπει οπωσδήποτε να το λύσουμε αν θέλουμε να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά σε αυτό το κλάδο. Επίσης ε, έχουμε παραγγείλει μία μελέτη και για τη φορολόγηση, μόνο για τους τοπικούς φόρους αλλά και γενικότερα για τους ε, φόρους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσει ε, στον τουρισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερο θέμα που απασχολεί την Επίτροπο. Και συμμεριζόμεθα πλήρω αυτά που είπατε για την συνδεσιμότητα. Η συνδεσιμότητα είναι η βάση για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες παντού στον τουρισμό. Για τη βιωσιμότητα. Η Επιτροπή, όπως ξέρετε, έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα δικτών για να ε, μετρήσουμε την ε, ε, εργασία που κάνουν οι διάφοροι φορείς για την βιωσιμότητα, ούτως ώστε να υπάρξουν και βραβεία στους προορισμούς που εφαρμόζουν καλύτερα αυτούς τους δείκτες. Αυτό το σύστημα δικτών είναι τώρα στη διάθεση όλων των ευρωπαϊκών προορισμών. Θα το τροφοδοτήσουμε, θα στηρίξουμε τη λειτουργία του, αλλά οι ίδιοι οι προορισμοί πρέπει να συνεργαστούν με φυσικά όλη μας τη στήριξη. Βιωσιμότητα, όπως υπόθηκε από έναν Ευρωβουλευτή, είναι θέμα και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και θέμα αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά, το σχέδιο Juncker μπορεί να βοηθήσει πολλές ε, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για παράδειγμα να επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των εκπομπών. Αυτό θα βοηθήσει και τη βιωσιμότητα, αλλά και τα περιθώρια κερδοφορίας τους σε, μια, σε ένα κλάδο που έχει προβλήματα με το επίπεδο κερδοφορίας του. Για τη στρατηγική. Ήρθε εδώ η Επιτροπός μου, άρα δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που σας είπε. Προσπαθούμε να εκπονήσουμε τώρα ένα πρόγραμμα δράσης που θα προσπαθήσει να προωθήσει τις προφανείς και σημαντικές ε, ε, προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ του τουρισμού και των πολιτιστικών και δημιουργικών προσπαθειών και εγχειρημάτων. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και σας ευχαριστώ θερμός. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα για να κλείσει ο Ισανίου Βουέι, ο πρόεδρος ε, της Ομάδας Εργασίας για τον Τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή ανταλλαγή. Καμιά φορά επικρίνω κι εγώ ε, την πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι συχνά οι ευρωβουλευτές ε, μιλούν για μεγάλα επίβολα σχέδια και ακούμε μεγάλα λόγια που δεν γίνονται ποτέ πραγματικότητα. Τώρα όμως ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το τελευταίο χρόνο και παραπάνω συνεργάζομαι με τους συναδέλφους για το μανιφέστο αυτό ε, τη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας και με παρακάλεσαν να ε, παίξω ένα ρόλο διαμεσολαβητικό. Να δούμε πώς θα συνδέσουμε την πολιτική με τον κλάδο και τα τουριστικά επαγγέλματα. Έχω διάφορες συστάσεις ε, και θα πρότεινα να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με αποδέκτες τον Επίτροπο Ναύρατσης και τις ε, κρατικές αρχές. Δεν θα πρέπει ο, ο τουρισμός ε, να ε, γίνει ένα μάθημα στο σχολείο. Σε περισσότερα κράτη-μέλη δεν διδάσκεται ο τουρισμό στα σχολεία. Εμεί υποστηρίζουμε πολλά προγράμματα σπουδών κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι μάθημα στο σχολείο. Επίση, σε ό,τι αφορά τι στατιστικέ και τι διάφορε κατηγορίε και του δείκτε για να μετρούμε ε, τις θέσεις εργασίας, ε, τα έσοδα που προκύπτουν κτλ. Συμφωνώ και με τον κύριο Νίλσον για το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιμέρους επιτροπών στο Κοινοβούλιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και θα προσπαθήσουμε μαζί με άλλους ε, Συναδέλφου τη Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής να κάνουμε μια μελέτη την οποία θα μπορούμε όλοι να χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο της Επιτροπής και όλα τα μέλη που μίλησαν. Ε, παρακαλώ να μας βοηθήσετε για να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη επιτροπή στην οποία θα πρέπει να αποταθούμε, Επιτροπή Εσωτερικών, ΛΥΜΠΕ, ε, θα μπορούσε να δημοσιεύσει ε, μία ανακοίνωση για το πρόβλημα θεωρήσεων διαβατηρίων για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Συγκεκριμένα, ας πούμε, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μπορούσε να επιληφθεί και ε, να συνεργαστεί μαζί μας για την κοινή μας προσπάθεια, γιατί μας απασχολεί και μας το θέμα. Στη συνεδρίαση των συντονιστών αναφέραμε αυτό το θέμα και θα ε, φροντίσουμε να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή Ελευθεριών. Και κάτι άλλο που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ε, το οικονομικό ζήτημα. Θα πρέπει να έχουμε τον προπολογισμό ε, για την υπηρεσία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το τμήμα που ασχολείται με τον τουρισμό, χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δραστηριότητα και η λειτουργία αυτής της μονάδας και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Και τελευταίο που θέλω να σας αναφέρω είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ακούστηκε, τουριστική ε, πρωτεύουσα. Ε, η υπόθεση αυτή μας απασχόλησε στην ομάδα του Μανιφέστο και με τον κύριο Σανταντέρ και με άλλους. Θα μπορούσε να είναι μια κοινή πρωτοβουλία ε, του κλάδου και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γιατί να μην λανσάρουμε την ευρωπαϊκή τουριστική πρωτεύουσα. Ε, είναι ε, μια καλή πρόταση και ο κύριος Κοράτζα για υπηρεσίες του στο τμήμα του πρόσφατα έκαναν μια σχετική εκδήλωση με παρουσία τριών επιτρόπων όπως ακούσαμε. Οι τρεις επίτροποι λοιπόν ε, δήλωσαν και οι τρεις ε, ότι υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και με τον κύριο Ναύρατσης ε, έχω διοργανώσει μια εκδήλωση για τα μέλη που συνέταξαν το μανιφέστο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία, Ευρωπαϊκή Τουριστική Πρωτεύουσα, γιατί όχι, πάρα πολύ καλή πρόταση και θα μπορούσε να υποστηριχθεί από δεξιούς αριστερούς μέχρι και τους πρασίνους μπορούμε να πείσουμε να μας υποστηρίξουν, φανταστείτε, και άλλες πολιτικές ομάδες. Και νομίζω ότι στην παρούσα θητεία ε, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και θα ήταν σημαντικό επίτευγμα και κατάκτηση. Να έχουμε κάθε χρόνο στην Ευρώπη, εκτός από την πολιτιστική και μια τουριστική πρωτεύουσα και με οικονομική αντίστοιχα στήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Η Ούρσουλα και εγώ συμφωνήσαμε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό σε κάποια επόμενη συνεδρίαση της Task Force να ε, κάνουμε μία ε, απογραφή όλων των ταμείων ε, που δίνουν κονδύλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντληθούν πόροι για την ενίσχυση του τουρισμού, για να έχουμε έτσι μια γενική εικόνα, μια επισκόπηση όλων αυτών των διαθέσιμων πόρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση και την υποστηρίζω. Και μια τελευταία παρατήρηση. Αύριο το βράδυ έχουμε και μία ακόμα σημαντική εκδήλωση και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Περί τίνος πρόκειται. Έχουμε μια σύνοευρωπαϊκή συνεργασία στο τομέα του τουρισμού. Έχουμε βρει ένα νέο τρόπο συνεργασίας με τους Κινέζους, για την οποία θα συζητήσουμε αύριο το άλλο Σανταντέρ και άλλοι ε, συμμετείχαν ε, στη διοργάνωση αυτή για τη συνεργασία Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος ενδιαφέρεται, ε, είστε προσκεκλημένοι και σας περιμένουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρουσιάσεις σας και για τη συμμετοχή σας. Για όλους όσοι συνεισέφεραν στην οργάνωση και ευχαριστώ και τους μεταφραστές που μας έδωσαν 10 λεπτά παραπάνω υπέρβαση ωραρίου. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και εδώ ολοκληρώνεται η πρωινή μας συνεδρίαση. Να πάτε στο καλό.